Ωραία. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ καθίστε. Σας ε, καλωσορίζω στην ε, συνεδρίαση αυτή της Επιτροπής μας. Έχω την τιμή να προεδρεύω ως προσωρινή πρόεδρος, ως πρώτη, απερχο... πρώτη απερχόμενη αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1, το οποίο ισχύει τις μουτάντης και για τις ε, συνεδριάσεις επιτροπών. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής μας ε, και άρχεται η συνεδρίαση. Ο στόχος της ε, σημερινής μας συνεδρίασης είναι να εκλέξουμε το Προεδρείο τον, ή την Πρόεδρο και μέχρι τέσσερις αντιπροέδρους της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 204 του κανονισμού. Πρώτα απ' όλα λοιπόν εκλέγουμε τον ή την Πρόεδρο, μετά αντιπροέδρους. Επίσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε εάν έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Εάν δεν τις έχετε παρακαλώ ζητήστε αμέσως μία ε, άλλη κάρτα, αλλιώ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορία. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο, αλλά εάν χρειαστεί κάτι τέτοιο θα χρειαστείτε την κάρτα ψηφοφορία. Σύμφωνα με το άρθρο 200 του κανονισμού ανακοινώνω πώς ε, λαμβάνουν μέρος τα εξή αναπληρωματικά μέλη στην ψηφοφορία και θα σα πω και ποιο αντικαθιστά ποιον. Ο κύριο Άξελ Φω αντικαθιστά τον κύριο Καλχαιντ Μπέκερ, ο κύριος Κοέλιο αντικαθιστά την κυρία Μαντέρα. Ο κύριος Στέτινα αντικαθιστά την κυρία Μουσολίνη. Η κυρία Σλάιν αντικαθιστά την κυρία Φλασίκο Βαμπένοβα. Ο κύριος Φερνάντες αντικαθιστά τον κύριο Λόπεζ Αγγιάρ. Ο κύριος Γιούρεκ αντικαθιστά τον κύριο Τομασεύσκη. Η κυρία Κάλλας αντικαθιστά την κυρία Γκρίσμπεκ. κυρία Βίρινγκ αντικαθιστά τον κύριο Μισελ, η κυρία Σπινέλη αντικαθιστά την κυρία Αστ και η κυρία Λούνατσεκ αντικαθιστά την κυρία Βαλέρο. Αυτοί λοιπόν είναι οι αναπληρωτές και θα ήθελα να πω πως θα πρέπει οι πολιτικές ομάδες να ενημερώσουν για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά τα οποία ανέφερα πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ερχόμαστε τώρα στην εκλογή Προέδρου. Όσον αφορά την Ολομέλεια, την ε, μισή απαρτία, βλέπω πως υπάρχουν πάνω από 15 βουλευτές παρόντες, οπότε έχουμε απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 208 παράγραφος 2. Και τώρα περνάμε στις υποψηφιότητες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν υπάρχουν υποψήφοι για την θέση του Πρόεδρου, κυρία Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω τον Κλοντ Μόραες να συνεχίσει ως πρόεδρος της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής ο υποψήφιος, όπως είναι ο κύριος Μωραές, και να έχει υποβάλει και την δήλωση οικονομικών συμφερόντων, όπως έχει κάνει ο κύριος Μωραές. Έχουμε λοιπόν υποψήφιο τον κύριο Μωραές. Κλοντ, δέχεστε την υποψηφιότητα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα. Περνάμε στην ψηφοφορία. Ένας είναι ο υποψήφιος. Οπότε προτείνω να γίνει εκλογή Προέδρου διαβοής. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για την εκλογή του κ. Μωρέσ και τον παρακαλώ να αναλάβει την Προεδρία. I have Μεταξύ να σας εξομολογηθώ πως αν προταθώ ως αντιπρόεδρος θα είμαι το μέλος αυτό το οποίο θα έχει την μακρότερη συνεχή θητεία στο Προεδρείο από το 2007. That was a relief. Thank you. Τι ανακούφιση. Ευχαριστώ, Κίνγκα. Πριν περάσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους και για τις εργότερες προσπάθειες που καταλάβαμε την τελευταία διετία. Γίναμε αυτό που γίναμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών χάρη στην ενεργό δράση των ε, μελών της Επιτροπής τώρα πια μα θεωρούν πολύ δραστήρια και πολύ απασχολημένη, φορτωμένη επιτροπή. Χάρη στην σκληρή προσπάθεια που κάναμε και στα επιτεύγματά μας τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Και είναι μεγάλο προνόμιο για μένα η επανεκλογή μου και σας υπόσχομαι ότι θα εργαστώ ακόμη πιο σκληρά και θα είμαι όσο πιο ανοιχτό και διαλεκτικός γίνεται στο υπόλοιπο ήμιση της κοινοβουλευτική μας θητεία. Και σε ευχαριστώ θερμά που με, με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας πάντα, <laughs> παρόλο που δεν φαίνεται να είχατε καλή επιλογή. Ευχαριστώ πάντως για την υποστήριξη. Περνάμε τώρα στην εκλογή των αντιπροέδρων. Με βάση το άρθρο 204 του ιστορικού κανονισμού, θα πρέπει, όπως είπε πριν και η Κίνγκα, να αναγγείλω πιο αναπληρωματικά μέλη λαμβάνουν μέρος στην ψηφοφορία. Πρώτο, ο κύριος Φως για το ΕΛΚ, Κοέλιο για το ΕΛΚ, Στετίνα για το ΕΛΚ, Σλάιν από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες, Φερνάντες από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Γιούρεκα από το ΕΣΥΑΡ. Βίρνεκ από τους Φιλελεύθερους, μάλλον Κάλλας, επίσης για τους φιλελεύθερους και η κυρία Σπινέλη τέλος από την ΚΟΕ και η κυρία Τσέκ για τους πρασίνους. Αυτή είναι η αναπληρωματική που θα ψηφίσουν σήμερα. Περνάμε τώρα στην εκλογή των αντιπροέδρων. Σε ό,τι αφορά την απαρτία, διαπιστώνω ότι έχουμε συγκεντρώσει την απαρτία γιατί πάνω από 15 μέλη είναι παρόντα στη συνεδρίαση. Τώρα, υποψηφιότητες για τις ε, θέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου αντιπροέδρου και τέταρτου αντιπροέδρου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, είτε μια πολιτική ομάδα μπορεί να υποβάλει υποψήφιο, είτε τουλάχιστον 5% των μελών τη Επιτροπή. Δηλαδή, τρία μέλη τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών μπορούν να υποβάλουν μια υποψηφιότητα. Επίση, ο υποψήφιο θα πρέπει να είναι τακτικό μέλο τη Επιτροπή και να έχει υποβάλει δεόντω τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Παρακαλώ τους υποψηφίους ε, να δηλώσουν αν δέχονται την υποψηφιότητά τους. Πρώτος υποψήφιος, Βενσούλα. Ναι, θα θέλαμε να προτείνουμε την κυρία Κινγκαγκάλ για τη θέση της πρώτης αντιπρόεδρου. Μάλιστα, η κυρία Κινγκαγκάλ είναι υποψήφια για την πρώτη αντιπροεδρία. Άλλος κανείς για τη θέση αυτή, όχι. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, μπορούμε να ψηφίσουμε διαβοής την πρώτη αντιπρόεδρο. Διαβοής λοιπόν εκλέγουμε την κυρία Κίνκα Γκάλο, πρώτη αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Περνάμε στην εκλογή του δεύτερου αντιπρόεδρου. Ποιος είναι υποψήφιος? Κυρία Ζίπελ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα θυμάστε ότι ευτυχώς ή δυστυχώς χάσαμε την κυρία Γιώτοβα, οπότε προτείνω τον Σεργέη Στάνισεφ ως δεύτερο αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Κύριε Στάνισεφ, συμφωνείτε με την υποψηφιότητά σας, βεβαίως. Πρόκειται για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ξέχασα πριν να ρωτήσω την κυρία Γκάλα αν συμφωνούσε με την υποψηφιότητά της. Το εξέλαβα ως αυτονόητο. Πάντως συμφωνεί και ο κύριος Στάνισεφ. Οπότε κηρύσουμε την εκλογή του στη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Περνάμε στη θέση του τρίτου αντιπρόεδρου. My apologies, we didn't, um, Συγγνώμη, έπρεπε να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε διαβοή. Ε, συμφωνείτε με την εκλογή του κύριου Στανίσεφ για τη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Ωραία, περάμε στον τρίτο αντιπρόεδρο. Ποιο είναι υποψήφιο, η κυρία Σαρτζεντίνη, για να δηλώσει υποψηφιό... την υποψηφιότητα. Ναι, να δηλώσω την υποψηφιότητα εκ μέρου των Πρασίνων και για τρίτη συνεχή χρονιά τον κύριο ε, για, τη θέση του τρίτου αντιπροέδρου, τον κύριο Γιάνν Φίλιπ Άλμπρεχτ. Μάλιστα, ο κύριο Γιάνν Φίλιπ Άλμπρεχτ είναι ο τρίτο αντιπρόεδρο, υποψήφιο τουλάχιστον. Δεν υπάρχει άλλο κανεί υποψήφιο για τη θέση αυτή. Συμφωνεί με την υποψηφιότητα ο κύριο Άλμπρεχτ, οπότε να προσθέσουμε και τον κύριο Γιάνν Άλμπρεχτ. Ψηφίζουμε διαβοής πρώτα. και επιβεβαιώνουμε την εκλογή του. Κυρία Μετσόλα, να μας πει ποιος είναι υποψήφιος για την τέταρτη την Με χαρά και τιμή ε, θα θέλαμε να προτείνουμε την κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα για τη θέση της τετάρτης αντιπρόεδρου. Συμφωνείτε κυρία Κουντρίτσκα με την υποψηφιότητα. Ναι, άλλοι υποψήφοι δεν υπάρχουν. Οπότε πολύ ευχαριστώ να εκλέξουμε διαβοής και την κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα για τη θέση της τετάρτης αντιπρόεδρου. Um, να ζητήσω και από τους τέσσερις ε, αντιπρόεδρους μας να έρθουν στο Προεδρείο και θα διακόψουμε μέχρι τις 3.30 για να ξεκινήσουμε την τακτική μας ε, δημόσια συνεδρίαση. Μια μικρή διακοπή μέχρι τις 3.30 και στο μεταξύ να έχουν λάβει θέση οι αντιπρόεδροι στο Προεδρείο.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE Uh, Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε εγκαίρως. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει στην ημερήσια διάταξη, παρακαλώ λίγη ησυχία. Για το σημείο 6, την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη ο Γιάνν Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας εδώ δύο δικηγόρους που εκπροσωπούν τον Σνόντεν, ε, τον καταγγέλλοντα Σνόντεν και έχουμε και ένα ψήφισμα σχετικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου του 2015 που ζητούσε την προστασία των καταγγελόντων και ζητούσε από τα κράτη-μέλη να δώσουν άσυλο. Μήπως θα μπορούσαμε να δώσουμε λίγα λεφτά στους δύο αυτού δικηγόρους για να μας εξηγήσουν ποια είναι η κατάσταση με τη θέση του Σνόντεν. Ευχαριστώ, Γιάννη. Οι συνάδελφοι θα ξέρουν την παρουσία των δικηγόρων. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στο Κοινοβούλιο ε, όπου θα συμμετάσχουν αυτοί οι δύο δικηγόροι. Το αίτημα που κάνετε είναι να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να μας εξηγήσουν τις δραστηριότητες τους σε σχέση με το ψήφισμα το οποίο έχουμε ήδη ετοιμάσει. Προτείνω, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, συνάδελφοι, να ασχοληθούμε με το θέμα του συνόδου στο τέλος της συνεδρίας, αν μας επιτρέψει ο χρόνος. Το δέχονται, οι συνάδελφοι το δέχονται και οι δύο δικηγόροι. Ναι, κάνω ένα πρόβλημα. Ε, αν δεν υπάρχει, δεν δημιουργείται πρόβλημα, θα ήθελα και πριν να το κάνουμε. Αλλά εάν δεν μπορούμε, στο τέλος, εντάξει. Εντάξει, θα είμαι ευέλικτος. Και λέει ο πρόεδρος. Προς το τέλος της συνεδρίασης θα βάλουμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την ευελιξία σας στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, προχώρησε πολύ γρήγορα ε, και μαζί με τις ευχαριστίες μου είχα σαν σκοπό να ευχαριστήσω όλους ιδιωτέρως. Βέβαια, έχει συμβεί τώρα. Όλα τα μέλη που τακτικά συμμετείχαν, τους συντονιστές, τα μέλη της Επιτροπής που πάντα είναι παρόντα, αλλά και το προσωπικό. Το προσωπικό της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, τους ανώτατους υπαλλήλου που είναι πάντα εδώ και μας βοηθάνε. Και τα υπόλοιπα. Και τους υπαλλήλους βεβαίω των υπολείπων θεσμικών οργάνων όταν έρχονται βεβαίω. Και παρά την ένταση των εργασιών και τη δυσκολία της, των συνεδριάσεων της Επιτροπής, παρά τις πολιτικές δυσκολίες που έχουμε, ε, γινόμαστε λίγο-λίγο μια οικογένεια, χάρη στην πραγματογνωμοσύνη, χάρη στην, στο ζήλο των ανθρώπων ε, και την παρουσία τους εδώ, ε, και των ε, Ευρωβουλευτών, αλλά και των υπαλλήλων. Και των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίω των υπαλλήλων των άλλων θεσμικών οργάνων. Όλη αυτή μαζί, όλη αυτή η οικογένεια κατέστησε τη ΛΥΜΠΕ αυτή την επιτροπή την αναγνωρίσουμε που όλοι ξέρουμε σήμερα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν ε, τώρα στην ημερήσια διάταξη και ας περάσουμε στο σημείο 9 που είναι η κατάσταση της ένταξης των, όσον αφορά την ένταξη των Ρωμά στα κράτη-μέλη. Έχουμε θέσει το θέμα αυτό ε, που αφορά τα, την ισότητα και τα δικαιώματά τους σε πολλές φορές και είχαμε και ένα ψήφισμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα 2015. Σήμερα καλέσαμε τον κύριο Ιωάννη Δημητρακόπουλο, Διευθυντή του Τμήματο Ισότητα και Δικαιωμάτων του Πολίτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να μα παρουσιάσει τα απορίσματα τη δεύτερη έρευνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι Εθνικέ ε, Μειονότητε και τι Διακρίσει. Έχουμε και τον κύριο Σμιτ, ο οποίο ε, ε, διορίστηκε τμήματάρχη τη συντονιστική μονάδα στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη ε, θα ενημερώσουν τα μέλη της ΛΥΜΠΕ για την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για τους Ρωμά και τα επόμενα βήματα ε, στις πολιτικές για τους Ρωμά. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στον κύριο Δημητρακόπουλο και συνεχεία στον κύριο Σμιτ και συνεχεία θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ και τους δύο που ήρθατε. Και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που καλέσατε την υπηρεσία των Οργανισμών Θεμελιών Δικαιωμάτων να σας παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών του. Στοιχεία τα οποία δείχνουν τι σημαίνει να είσαι σήμερα Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2008, ο Οργανισμός Θεμελιών Δικαιωμάτων ετοίμασε την πρώτη έρευνα με τα στοιχεία με βάση τον πρώτο γύρο Ε, ερωτήσεων ε, για θέματα εθνοτικών μειονοτήτων και διακρίσεις και η εικόνα ήταν ζωφερή. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, το Συμβούλιο, ε, εξέδωσαν ψηφίσματα, πολιτικές πλαίσιο, συστάσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Εμείς κάναμε μια πιο στοχευμένη έρευνα το 2011 η οποία αφορούσε τέσσερις πτυχές της κοινωνικής ζωής ε, με λεπτομέρειες, δηλαδή ε, μπήκαμε σε περισσότερες λεπτομέρειες στα θέματα των διακρίσεων, κάνοντας συγκρίσεις για τη ζωή των Ρωμά σε σχέση με άλλες κοινότητες, τους γειτονέ τους. Και τώρα σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δεύτερη, του δεύτερου του τμήματος ε, ευρείας έρευνας, όπου συγκρίνουμε ε, την κατάσταση των Ρωμά σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό για να δούμε ότι μετά τις πολλαπλές προσπάθειες που έχουμε κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ρωμά, πόσο μακριά φτάσαμε. Τα αποτελέσματα, όπως βλέπετε στην έκθεσή μας, ε, συγκρίνονται με τις συστάσεις του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013 ε, και με τους, τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ για να δούμε σε ποιο βαθμό η προσπάθεια ένταξης των Ρωμά υλοποιούν αυτούς τους σημαντικούς διεθνείς στόχους. Τώρα, να σας πω δύο πράγματα για την έρευνα. Η έρευνα αυτή καλύπτει ε, τους Ρωμά σε νέα κράτη-μέλη, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτοκαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ισπανία. Καλύπτει περίπου 80 με 85% τον του πληθυσμού των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τι εκτιμήσει του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε περίπου 8.000 άμεσε συνεντεύξει, 45 λεπτών η καθεμία, όπου οι ίδιοι οι Ρωμά παρουσιάστηκαν ε, και δίνουν στοιχεία, δίνει στοιχεία αυτή η έρευνα για περίπου 34.000 νοικοκυριά και τα μέλη τους. Ο τρόπος ε, που κάναμε αυτή την δειγματοληψία ήταν ε, ένα τυχαίο μοντέλο και μια διοικητική μονάδα με τουλάχιστον 5 με 10% Ρωμά στο συνολικό πληθυσμό. Δηλαδή δεν πήγαμε απλώς ε, σε καταβλισμούς Ρωμά, έτσι μόνο και μόνο για να διευκολύνουμε τη ζωή μας, όπου συγκεντρώνονται κυρίως οι Ρωμά, αλλά προσπαθήσαμε να πάμε σε διοικητικές μονάδες, ας πούμε, των κρατών μελών ή περιοχές, ας πούμε, όπου δεν ζουν μόνο Ρωμά. Τα αποτελέσματα όμως είναι εξίσου αποθαρρυντικά με το παρελθόν. Κατά μέσο όρο, σε διαφορετικές χώρες, με, διαφορετικές, με πολύ μεγάλες διαφορές, δεν θέλω να μπω όμως τώρα σε λεπτομέρειε, δεν έχω το χρόνο. Φαίνεται ότι η μεγάλη πλειοψηφία, το 80%, ζουν κάτω από το κατόφλι κινδύνου φτώχεια ε, στη χώρα τους. Ε, ο ένας στους τέσσερι Ρωμά και πολύ πιο σημαντικό. Το ένα στα τρία παιδιά ε, πεινάνε τουλάχιστον μία φορά το μήνα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, αυτό πριν την έρευνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί για τα παιδιά όλα τα κράτη-μέλη ε, υπέγραψαν ε, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών και επιπλέον το άρθρο 33 της δικής μας συνθήκη λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών και να προωθήσει τα δικαιώματά τους. Τώρα, πού ζουν αυτά τα παιδιά και οι ενήλικες. Είδαμε τα σπίτια, τη στέγη. Ε, υπάρχουν πολύ, πολύ μεγάλα προβλήματα, ε, δεν υπάρχουν αρκετά επαρκή στέγη. Ο ένας στους τρεις Ρωμά ε, ζει σε σπίτι το οποίο δεν έχει τρεχόμενο νερό. Ένας από τους, στους δέκα ε, ζει σε σπίτι που δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα επιπλέον. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι για την εκπαίδευση έχουμε πρόβλημα. Ε, τα αποτελέσματα δείχνουν τεράστιες διαφορές, κυρίως σε, στη στέγη μεταξύ των Ρωμά και του υπόλοιπου πληθυσμού της χώρας ε, για την οποία ερευνήσαμε. Ένα άλλο ε, επιβαρυντικό στοιχείο είναι η πρόσβαση ε, στις υπηρεσίες κοινό ωφελίας. Το να έχεις επίσης ντους, μπάνιο, καζανάκι στο σπίτι κτλ. Και συχνά οι Ρωμά τελικά ζουν σε τεμάχια της γης, ας πούμε, ε, χωρίς ρυθμίσεις, ε, με, χωρίς βασικές, ε, οι βασικές ανάγκες δεν καλύπτονται. Τώρα, στον εκπαίδευση. Εδώ είναι το μέσο όπου μικρές βελτιώσεις έχουν εντοπιστεί, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά την ηλικία στην οποία ξεκινάνε τα παιδιά το σχολείο. Μόνο το 50% των παιδιών του Ρωμά ε, που ε, ελέγξαμε ας πούμε πάντα στο σχολείο ε, και μόνο το μισό των ε, Ρωμά πάνε στο Λύκειο. Επομένως, το θέμα των κοινωνικών δικαιωμάτων και το θέμα της ανεργίας των νέων όταν το συζητάμε, το γεγονός ότι δεν πάνε στο Λύκειο δείχνει ότι τους λείπει ένα βασικό εργαλείο για να βρουν δουλειά εν συνεχεία στην αγορά εργασία. Και τέλος, το 95% σχεδόν όλοι δεν πηγαίνουν ε, στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια τεχνική ανώτερη σχολή. Και παρά την νομική απαγόρευση που υπάρχει για, για την απομόνωση στα σχολεία, ε, η απομόνωση στα σχολεία ή εκ των πραγμάτων απομόνωση λόγω του τόπου όπου ζουν είναι πρόβλημα στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία. Μίλησα για την νεολαία. Τώρα, θα σας δώσω λίγα νούμερα τα οποία τονίζουν αυτό που είπα πριν. Κατά μέσο όρο, το 63% των νεαρών Ρωμά, 16 με 24 χρονών, ε, δεν δουλεύουν, δεν ε, λαμβάνουν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση σε σχέση με το 10% των συνομιλίκων τους που δεν είναι Ρωμά στις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεράστια η διαφορά αυτή, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί κάπως. Επίσης, να προσθέσω ότι... Τα αποτελέσματα δείχνουν και χάσμα μεταξύ των δύο φύλων. Κατά μέσο όρο 72% των γυναικών Ρωμά 16-24 ετών δεν ε, δουλεύουν ούτε εκπαιδεύονται σε σύγκριση με το 55% των ε, νεαρών γυναικών. Βεβαίως είναι ε, δύο κακές περιπτώσεις ε, και βεβαίως ε, αυτό το κενό είναι μεγαλύτερο σε Ελλάδα, Πορτογαλία και Ουγγαρία. Στο τα νούμερα για την Ελλάδα. 81% των γυναικών Ρωμά μεταξύ 16 και 24 ούτε εργάζονται ούτε εκπαιδεύονται. Όταν δούμε την απασχόληση για τον συνολικό πληθυσμό βλέπουμε ότι λιγότερο από... Λιγότερο από ένα στους τρεις απασχολούνται, 44% ζουν σε νοικοκυριά τα οποία χαρακτηρίζονται χαμηλής έντασης εργασίας, δηλαδή κάτω από το 20% της δυνατότητας του νοικοκυριού και καμιά φορά κάνουν δουλειές που πληρώνονται άσχημα και επικίνδυνες δουλειές όπως βλέπετε στη φωτογραφία όπως αυτή η γυναίκα η οποία προσπαθεί να βρει μέταλλα σε χωματερή και βεβαίως απασχόληση από αυτούς τους όρους Ε, είναι κάτι το οποίο περισσότερο από εμάς θα θεωρούσαμε απαράδεκτο. Και πάλι η συζήτηση για την ασφάλεια στην εργασία πρέπει να περιλαμβάνει και παραδείγματα Ρωμά που δουλεύουν υπό τέτοιε συνθήκες. Λοιπόν, όταν μιλάμε για διακριτική μεταχείριση, ε, βεβαίως αναφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα μέσα στην έκθεση, ο τίτλος, που νομίζω υπογραμμίζει την κατάσταση είναι ότι ζουν στο περιθώριο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. 41% θεωρούν ότι υφίστανται διακρίσεις στην κοινωνική ζωή και ιδιαίτερα θα τόνιζα παρά το ότι τα νούμερα δεν είναι ε, τόσο κοντά όταν έρχονται σε επαφή με την δημόσια διοίκηση όταν μπαίνουν σε ένα μαγαζί ή σε επαφή με τους ε, συμπολίτες τους 16 χρόνια μετά από την ε, υιοθέτηση της οδηγίας περί φιλετικής ισότητας μόνο 12%, 12 είπαν ότι θεωρούν ότι είχαν ε, υποστεί ε, κάποια διακριτική μεταχείριση και το ανέφεραν στις αρχές. Και επιπλέον όταν τους ρωτήσαμε αν γνωρίζουν την υφιστάμενη νομοθεσία, μόνο 36% γνώριζαν ότι υπάρχει τέτοια νομοθεσία κατά των διακρίσεων και 82% δεν ήξεραν κάποιο οργάνωση η οποία προσφέρει στήριξη σε τέτοια θύματα. Το άρθρο 10 της Οδηγίας ε, Περιφυλετικής Ισότητας μιλάει για την διάδοση πληροφοριών και λέει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να φροντίσουν οι διατάξεις οδηγίας αυτής να φτάσουν στα άτομα τα οποία αφορούν στην επικράτειά τους. Νομίζω λοιπόν πως η εφαρμογή της οδηγίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξαναδούμε υπό το φως των ευρημάτων αυτών. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω όπως έκανε και ο διευθυντής μας όταν παρουσίασε τα αποτελέσματα αυτά πέρσι τον Νοέμβριο, πως το θέμα αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι στόχη πολιτικής, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας, αφορά την ε, αξιοπρέπεια όλων των πολιτών της Ένωσης, ε, οποιαδήποτε καταγωγή και αν έχουν, και άρα σας παρακαλούμε ως ε, πολιτικοί να χρησιμοποιήσετε όλα τα δεδομένα που σας δίνουμε για να είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική που χαράζετε και πρέπει να αντιμετωπιστεί η αντίσταση στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής και πρέπει να καταπολεμηθεί η ε, τσιγκανοφοβία στην εφαρμογή της ε, πολιτικής και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων και τελειώνω με μία λέξη. Ενδυνάμωση τον Ρωμά, οι οποίοι πρέπει και οι ίδιοι να ασχοληθούν με το ζήτημα της ένταξής τους και βεβαίως σε συνεργασία με όσους θα ήθελαν να τους στηρίξουν. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ο κύριος Σμιτ θα ήθελα τώρα να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, όχι παραπάνω από ένα δεκάλεπτο, γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία και στους συναδέλφους να υποβάλουν διεξοδικές και αναλυτικές ερωτήσεις, γιατί είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι μερικοί συνάδελφοι με αυτό το θέμα. Οπότε, ένα δεκάλεπτο το πολύ για να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Σας περιμένει πληθώρα πολύ αναλυτικών ερωτήσεων. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επανεκλογή σας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τηρήσω αυτό το δεκάλεπτο που μου δώσατε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών της θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω αυτό που βλέπουμε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση της κοινωνικής ένταξης στο Ρωμά. Όπως γνωρίζετε ήδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τακτική ενημέρωση ε, για το πώς εκτιμά την κατάσταση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο και η τελευταία έκθεση ε, υπευλήθη στις 27 Ιουνίου του 2016. Οπότε ήδη είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε σχολαστικά τα επιμέρους σημεία αυτής της έκθεσης. Τώρα θα σταθώ στα πιο σημαντικά σημεία, στα πιο κέρια σημεία αυτής της αξιολόγησης. Η έρευνα με την αξιολόγηση αφορά αφενός το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο σε διάφορους κλάδους ε, και οριζοντίως ε, σε νομικό επίπεδο αλλά και σε θέματα απασχόλησης υγείας, ε, στέγασης καθώς και διαρθρωτικά μέτρα και μέτρα χρηματοδότησης. Επιπλέον, στη φετινή μας έκθεση στην Περσίνη ουσιαστικά, γιατί ήταν το 2016, για πρώτη φορά έχουμε ε, πίνακες και δελτία για κάθε ε, επιμέρους χώρα, με πιο αναλυτικές πληροφορίες και αξιολόγηση για την κάθε χώρα. Αυτό που ενδιαφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα θετικά σημεία, και είναι σημαντικό να τα επισημάνουμε. Έχουμε ήδη τις δομές ε, για το συντονισμό, για την ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών και για την παρακολούθηση της κατάστασης. Έχουμε το δίκτυο των ε, σημείων επαφής για τους Ρωμά. Τέτοια ε, σημεία επαφής υπάρχουν σε όλα τα κράτη-μέλη, οπότε οι αρμόδιες αρχέ κάθε χώρα ευρωπαϊκής Ένωση συγκεντρώνουν πληροφορίες και στα πλαίσια του δικτύου αυτού συζητούν τα θέματα και ανταλλάσσουν τι καλύτερε πρακτικέ. Επίσης, έχουμε και συναντήσεις κοινωνίας των πολιτών στα κρατη πέραν των συναντήσεων των αρμόδιων αρχών. Έχουμε ένα διτό σύστημα, ε, δύο επιπέδων. Έχουμε τις εθνικές πλατφόρμες Ρωμά στα κράτη-μέλη που λειτουργούν καλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά πολύ σημαντικές αυτές οι πλατφόρμες, αυτά τα δύο επίπεδα, για την ανταλλαγή πληροφοριών και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών και με τις ε, κυβερνήσεις, με τις διοικητικές δομές. Και είναι πολύ σημαντικό και το επισημαίνουμε τρεις φορές ότι έχουμε αυτή τη στιγμή σαφή σύνθεσμο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την ένταξη των Ρωμά, την κοινωνική του ένταξη, με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Κάτι που δείχνει και απτά ότι ήδη από το 2013 έχουμε στις ε, ειδικέ συστάσεις αναχώρα ειδικέ συστάσεις προς τα κράτη-μέλη που υστερούν κάπως ε, ακόμη στο θέμα της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Και τους ευχαριστούμε την προσοχή στο σημείο αυτό. Πολύ σημαντικούς μηχανισμούς λοιπόν έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης έχουμε και το θέμα της ε, χρηματοδοτικής υποστήριξης, της οικονομικής ενίσχυσης και στα κράτη-μέλη όπου οι ειδικές συστάσεις αναχώρα ισχύουν, έχουμε και την κοινωνική ένταξη των Ρωμά πλήρως ενσωματωμένη στα προγράμματα χρηματοδότησης. Και μιλούμε για προγράμματα 1,5 δις συνολικά ευρώ που δίνουν τεράστιες ε, δυνατότητες στα κράτη-μέλη για άντληση κονδυλίων. Επίσης, έχουμε ειδικά προγράμματα, ειδικώ αφοσιωμένα στους Ρωμά, ειδικώ αφιερωμένα στους Ρωμά, τα οποία δρομολογούμε απευθείας από τις Βρυξέλλες. Το πρώτο είναι ένα που ξεκίνησε πέρυσι, από τους ε, Ρωμά, για τους Ρωμά, για την αδελφοποίηση πόλεων, πολιτισμικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, ε, αφύπνιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνειδητοποίηση του θέματος. Και επίσης έχουμε και ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων για τα δικαιώματα των πολιτών και την ισότητα μεταξύ των πολιτών. Και εκεί έχουμε πολλές οργανώσεις Ρωμά που είναι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος επιχορηγήσεων και συμμετέχουν σε αυτό. Και τέλος, ε, πολύ σημαντικό είναι και το νομοθετικό επίπεδο γνωρίζετε τις δύο πολύ σημαντικές ε, ε, οδηγίες που ισχύουν, την οδηγία για την ε, φιλετική ισότητα και την απόφαση πλαίσιο του, Συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Επίσης, θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό να επισημάνω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει, ειδικά την τελευταία διετία, να εγκύπτει εις βάθος και στις έμπρακτες ε, εφαρμογές αυτές της νομοθεσίας. Και μάλιστα μερικές φορές κινήσαμε και τη διαδικασία επιπαραβάση, επιβολής κυρώσεων όταν διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται μόνο με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Οπότε, αυτό που θα ήθελα να επισημάνω από την έκθεσή μας δεν είναι να δώσω την εντύπωση ότι είμαστε συγκαταβατικοί ή αυτάρεσκοι. Απλώς θα πρέπει να επισημάνω ότι οι βασικές αυτές οι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω επιτυχία, αυτές οι δομές υπάρχουν. Δεν είναι λοιπόν καμία συγκατάβαση από μέρου μα. Και το θέμα είναι να δούμε τι επιτυχάνουμε επιτόπου, τι βιωτικέ συνθήκε, κατά πόσο οι συνθήκε διαβίωση βελτιώνονται για τον πληθυσμό των Ρωμά. Και σα παραπέμπω στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δυστυχώς ε, δεν μας έχει παρουσιάσει και πολλά θετικά σημεία. Μόνο δύο στοιχεία ε, τραβούν την προσοχή μου και που είναι κάπως πιο ελπιδοφόρα ως προς την κατεύθυνση που ακολουθούμε. Το πρώτο είναι, και μην με παρεξηγείτε, αλλά ένα από τα θετικά σημεία είναι ότι το ποσοστό φτώχειας είναι 80%. Βέβαια δεν είναι θετικό αν το δει κανείς απόλυτα, γιατί Ποιος ε, μπορεί να συμφωνήσει με ένα τόσο υψηλό ποσοστό φτωχών. Αλλά πριν από μία πενταετία ήταν 90% αυτό το ποσοστό. Απίστευτο και όμω αληθινό. 90% πριν από μία πενταετία το Ρωμά ήταν στο κατόφλι της φτώχεια. Και ακόμη και με την αργή αυτή ταχύτητα σημειώνουμε κάποια πρόοδα, αλλά απλώς θα πρέπει να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Αυτή ήταν μια πολύ μετριοπαθής ε, κατάσταση, ένα πολύ μέτριος δείκτης. Κάτι που είναι πιο ενθαρρυντικό είναι η ε, προσχολική εκπαίδευση. Ξέρουμε όλοι ότι η παιδεία είναι το κλειδί της καλύτερης κοινωνικής ένταξης. Και ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία η εκπαίδευση σε αυτή τη φάση είναι πολύ σημαντική. Και εδώ είναι ο μόνος τομέας που διαπιστώνουμε ότι η ένταξη των παιδιών άσχετα με την εθνοτική του καταγωγή βελτιώνεται σε μερικά κράτη-μέλη τουλάχιστον και για τα παιδιά Ρωμά είναι πάνω από 90%. Τέτοιου είδους δείκτες χρειαζόμαστε που είναι πολύ ενθαρρυντικοί και μακάρι τόσο ενθαρρυντικοί να ήταν και στα άλλα ε, επιμέρους τμήματα της μελέτης. Πάντως σίγουρα η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, το αντίθετο. Στην έκθεση έχουμε και κάποιες συστάσεις η πρωταρχική αφορά την εφαρμογή της ισχύωσης νομοθεσίας. Η εφαρμογή της οδηγίας κατά του ρατσισμού και η εφαρμογή της απόφασης ε, πλαίσιο του Συμβουλίου. Επίσης, ε, εντοπίσαμε το συγκεκριμένο πρόβλημα των εξώσεων ε, των ε, μελών των εθνωτικών μειονοτήτων. Απαράδεκτο αυτό. Επίση, ε, επισημάναμε το πρόβλημα του σχολικού διαχωρισμού, της απομόνωσης, τη κοιτοποίησης των σχολείων, τα προβλήματα τη κατοικία, τη στέγαση και ζητήσαμε πιο οριζόντιο χαρακτήρα των παρεμβάσεων και εξορθολογισμό του, ώστε να φτάνουν αυτέ οι παρεμβάσει στου Ρωμά, ιδιαίτερα όταν ε, πρόκειται για κρατικά κονδύλια. Επίσης, θα πρέπει να βελτιώσουμε και τη μεθοδολογία μας στη συγκέντρωση των δεδομένων. Χρειαζόμαστε καλύτερους μηχανισμούς παρακολούθησης της κατάστασης. Αυτές είναι οι βασικές συστάσεις της έκθεσής μας. Θα ήθελα τώρα εν συντομία να σας δώσω και μία επισκόπηση των δράσεών μας από τα μέσα του 2016 μέχρι σήμερα. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει αμέριστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την έκκλησή του για αναγνώριση της ημέρας της μνήμης. Λάβαμε και εμείς ενεργά μέρος ε, στις εκδηλώσεις της Δευτέρα Αυγούστου για την ημέρα της μνήμης. Επίσης, ξεκίνησαν διάφορα πρόσθετα προγράμματα. Πάντως η πιο σημαντική υλοποίηση είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου, που τα κράτη-μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να αναλάβουν περαιτέρω δράσεις για πολλούς τομείς. Δεν πρόκειται να τους ε, ε, απαριθμίζω τώρα. Η αθηγανοφοβία, η αξιολόγηση του προβλήματος, Αυτές οι δεσμεύσει των κρατών μελών συνιστούν σημαντικότατο βήμα προόδου και είμαστε ιδιαίτερω υπερήφανοι που καταφέραμε αυτές τις δεσμεύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σε θέση με τις υπηρεσίες της ε, τώρα που έχουμε ξεπεράσει την ενδιάμεση αξιολόγηση, να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης όσο πιο ευρύ γίνεται, με συμμετοχή των ενδιαφερομένων και παρόλο που χρησιμοποιούμε και εξωτερικές αξιολογήσεις και έρευνες, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τεκμήρια, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε ακόμη στο σωστό δρόμο, αλλά θέλουμε τα ακριβή στοιχεία και τα τεκμήρια αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να συσπηρωθούμε, να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας και να ξεκινήσουμε έναν ευρύτατο απολογισμό. Ελάχιστα ξεπέρασα το δεκάλεπτο, 55 δευτερόλεπτα, συγχωρήστε με, μα σας ε, Ανέφερα το χρόνο και τον περιορισμό γιατί έχουμε πολλούς ευρωβουλευτές που εδώ και χρόνια ασχολούνται με το θέμα των Ρωμά από το 1999 ε, και το 2004 με τη μεγάλη διεύρυνση υπήρξε κάπως βελτίωση κατάστασης. Γι' αυτό και λέω να δώσουμε το λόγο στους ευρωβουλευτές που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με το θέμα για να υποβάλουν λεπτομεριακές ερωτήσεις. Είναι μακροσκελέστατος ο κατάλογος, Οπότε θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους ε, με τη σειρά που τον ζήτησαν. Θα ήθελα να ξεκινήσω εγώ με μια ερώτηση που αφορά κάτι που επισημάνατε και οι δύο. Γιατί και οι δύο αναφέρατε το νομοθετικό πλαίσιο, την οδηγία κατά του ρατσισμού και την ε, απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου. Και μάλιστα τα πιο παλιά μέλη της Επιτροπής θα θυμούνται ότι αυτά είναι τα δύο ε, νομοθετικά εργαλεία που συνιστούν το νομοθετικό πλαίσιο και υποτίθεται είναι εκεί για να προστατεύσουν τους Ρωμά. Οπότε, σας ερωτώ, θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και πραγματικά υλοποιεί το ρόλο του, δηλαδή να προστατεύει την ε, μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή, την πολυπληθέστερη μειονότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείτε ότι είναι αρκετά αυτά τα δύο νομοθετικά εργαλεία. Η οδηγία για τις κατά των φιλετικών διακρίσεων δεδομένη της περιπλοκότητας και της δυσκολίας του θέματος, γιατί η οδηγία για την φιλετική ισότητα είχε σχεδιαστεί πριν το 2004. Πριν δηλαδή γίνει λεπτομεριακή ανάλυση του ζητήματος των Ρωμά. Γιατί αναφερθήκατε στο νομοθετικό πλαίσιο. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει αυτό. Η Σοράγια είναι η πρώτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Eh, Είχαμε eh, την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων με πολύ ανησυχητικά στοιχεία, τρομακτικά θα έλεγα, ε, παρόλο που δεν μας ευνηδιάζουν, γιατί ενεργοποιούμε, δραστηριοποιούμε στο θέμα αυτό και είμαι ακτιβίστρια για χρόνια πολλά και στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ερωτώ, πώς φτάνετε στους Ρωμά που είναι δεσπαρμένοι, μερικοί μένουν και στα δάση. Ξέρω ότι οι καταβλισμοί υπάρχουν χιλιάδες και οικισμοί Ρωμά, που είναι μακριά από οποιαδήποτε πόλη, χωριό ή κοινότητα. Έχουμε από 500 μέχρι 1000 και κατοίκους σε τέτοιου είδους οικισμούς, χωρίς πρόσβαση στην επικοινωνία, δεν έχουν καν πόσιμο είδωρ. Είναι ε, εγκατασπαρμένοι αριστερά και δεξιά και είναι πολλοί Ρωμά που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Τους καλύψατε στην ε, έρευνά σας. Επίσης, ε, η ερώτησή μου αφορά την πρόοδο που μπορούμε να σημειώσουμε. Εκπονούμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για τους Ρωμά και προσβλέπω σε στενή συνεργασία και με τον ΦΡΑ, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ασχολούμαι 30 ολόκληρα χρόνια με το θέμα αυτό και διαπιστώνω ότι υπάρχει α, μερικές φορές κινησμός, αλλά η αναγνώριση και μόνο τη ύπαρξη στο Ρωμά είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά θέλουμε μεγαλύτερη δραστηριοποίηση υπέρ των Ρωμά, γιατί να μην έχουμε και μία πραγματική επιτροπή αλήθειας για να αποκατασταθεί η αλήθεια για το θέμα αυτό. Και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στην ανάλυση της κατάστασης σε τέσσερις τομείς. καλά τα θέματα της υγείας, της απασχόλησης, ε, της ε, στέγης, της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικοί αυτοί οι τέσσερις τομείς, αλλά υπάρχουν και άλλοι τομείς που ενδιαφέρουν. Χρειαζόμαστε μια πραγματική επιτροπή αλήθειας και επανασυμφιλίωσης για τους Ρωμά. Γιατί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο επέσχετες είναι αυτές οι διακρίσεις εις βάρος των Ρωμά, γιατί δεν θεωρούνται ε, και ντροπή τέτοιε διακρίσεις αυτή τη στιγμή ακόμη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό της κατάστασης και να δούμε ποια είναι τα ιστορικά αίτια που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε φυσικά τους στόχους μας αλλά αυτές οι διαδικασίες επί παραβάση που έχετε ξεκινήσει κατά της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας ε, και άλλων χωρών, σε τι στάδιο βρίσκονται και πώς θα προχωρήσετε από εκεί και πέρα. Τι γίνεται με τις διαδικασίες επί παραβάση κατά της Ελλάδος και της Ιταλίας ή και άλλων χωρών. Επίσης, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζουν ότι γίνονται αναγκαστικές εξώσεις Ρωμά στη Βουλγαρία. Θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα το ζήτημα των αναγκαστικών εξώσεων. Επίσης, ε, και το Περιφερειακό Ταμείο και τα Διαρθρωτικά Ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επανέλθουν οι Ρωμά στα σπίτια τους. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Κορνίλια Έρνστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Γιατί η μελέτη αυτή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όλα τα γεγονότα επιτάπτως και πραγματικά είναι θλιβερά και την εντύπωση ότι μεταχειριζόμαστε τη Ρωμά σαν ανθρώπου οι οποίοι κουβαλήθηκαν από κάπου, αλλά υπάρχουν, ζουν αιώνε στην Ευρώπη. Και το ερώτημα είναι πώ η στρατηγική που έχουμε είναι πραγματικά σωστή και επιτυχημένη. Και το ερώτημά μου είναι ότι το 2011 αποφασίσαμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωση για τη Ρωμά με πολλέ φανφάρε. και συχνά την αναφέρουμε. πώς θεωρεί η Κομισιόν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο σοβαρά μέτρα κατά των κρατών μελών για να τηρήσουν τα όσα πρέπει να κάνουν ή θεωρείτε ότι με τα μέτρα τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής ε, μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Επόμενο. Υπάρχει μία μελέτη για την ε, καταναγκαστική στήρωση ε, πριν από ένα μήνα δημοσιοποιήθηκε. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας. Τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν γι' αυτό. Ειδικά στην ε, Τσεχία έχουν σταματήσει οι καταναγκαστικές στηρώσεις ή συνεχίζονται ακόμα. Το ίδιο επίσης αφορά και την, ε, τα χωριστά σχολεία, καθώς πήγαιναν σε ειδικά σχολεία τα παιδιά των Ρωμά μαζί μάλλον με τα παιδιά με ειδικέ ε, ανάγκες. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ Κλοντ, ε, ανήκω σε αυτούς που ανέφερες, ε, ασχολούμαι με το ζήτημα εδώ και χρόνια και πραγματικά καλοδεχούμενη αυτή η έκθεση. Πραγματικά είναι πολύ ενισχυτικό αυτό. Οι Ρωμαίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους μας και είναι πολύ ενισχυτικό αυτό το οποίο είπατε για τα παιδιά. Το 2014 είχα αποβάλει μια ερώτηση προς την Κομισιόν και χαίρομαι που ακούω ότι η Κομισιόν θα αναλάβει να κάνει κάτι, γιατί προφανώς τα κράτη-μέλη δεν εφαρμόζουν την στρατηγική που είχαμε υιοθετήσει στην προηγούμενη θητεία και το ερώτημά μου προς την Κομισιόν ήταν πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το κοινωνικό ταμείο, το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης κτλ. Και η απάντηση που μου δώσαν ήταν ότι δεν μπορούσαν να εγγυηθούν αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ένταξη ε, και την ενσωμάτωση γιατί δεν ήταν αρκετά ισχυρή οι εθνικοί θεσμοί και δεν υπήρχε συντονισμός μεταξύ των εθνικών αρχών. Οπότε από το 2014 μέχρι σήμερα έχει υπάρξει κάποια βελτίωση. Ε, επισκέφθηκα μόνη μου το κράτος μέλος, ένα κράτος μέλος που έχει σοβαρά προβλήματα και δεν εντυπωσιάστηκα. Δεν υπάρχει ακόμα διαφάνεια για το πώς χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, να έχουν στέγαση και να μην υπάρχει γκαιτοποίηση. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν και πάλι τι θα γίνει για να διασφαλίσουμε ακριβώς ε, την δημιουργία ικανοτήτων στην διοίκηση και την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τέλος, για τα δελτία ταυτότητας. Γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα, ειδικά για τα παιδιά για την πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες ε, και τα σχολεία, όπως σωστά επισημάνατε, που σχετίζονται με το ότι δεν υπάρχει καν ε, ταυτοποίηση, δεν έχουν χαρτιά. Όταν λέω για ταυτότητα, ε, ε ενώ να αναγνωρίζονται ως πολίτες που έχουν πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ο αποκλεισμός έχει φτάσει σε τέτοιε διαστάσεις. Υπάρχουν χιλιάδες Ρωμά που θεωρούν ότι εξαναγκάζονται de facto να φύγουν από τη χώρα τους και πάνε σε άλλες χώρες με ακόμη χειρότερες συνθήκες. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά οξύτατη και ελπίζω να γίνει κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πίτερ Νιντερμίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έρευνά σας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βέβαια μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για την μεθοδολογία και πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους ε, τσιγκάνους κτλ. Μια άλλη στιγμή όμως. Να αφαιρθώ λίγο στις πολιτικές συνέπειες. Γιατί έχω καμιά φορά την ε, εντύπωση ότι είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές σε διασκέψεις, συναντήσεις, ε, διακηρύξει και στην πραγματικότητα τίποτα δεν συμβαίνει. Ε, έχω λοιπόν δύο πολύ σημαντικά πράγματα που θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι αισιόδοξο για την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων που αναφέρατε, καθώς ε, η εμπειρία μου από τη δική μου χώρα και από άλλες χώρες είναι ότι έχουμε θεσμικά όργανα κτλ. Αλλά τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν λοιπόν επ' αυτού. Ποιες είναι οι πολιτικές δυνατότητες άσκησης πίεσης πρώτον. Δεύτερον, βεβαίω ο ρόλος ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών, γιατί η εμπειρία μου είναι ότι πολλές ΜΚΟ είναι πολύ δραστήριες ε, επιτόπου στις τοπικές κοινότητες και γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που επιτίθενται σε αυτές τις ΜΚΟ. Έχουμε λοιπόν κάποιες δυνατότητες και υποχρέωση θα έλεγα να αλλάξει η κατάσταση και να συνεργαστούμε στενότερα με τις ε, οργανώσεις αυτές της ε, κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε πως η Κομισιόν ε, παίζει ρόλο εφαρμογή της νομοθεσίας με πολλούς τρόπους. Πρέπει λοιπόν να απαντηθεί το ερώτημα. Τι περισσότερο μπορείτε να κάνετε, γιατί τελικά είναι υπόθεση των ε, κρατών μελών. Νομίζω πως άκουσαν κάποιες ιδέες σήμερα. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ. Για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και για την καταγγελία μιας κατάστασης η οποία είναι αποθαρρυντική. Στην έκθεση κάνετε λόγο για σοβαρότατες ελλείψεις ε, απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Νομίζω ότι η λύση βρίσκεται στο να ενισχύσουμε την κοινότητα τρόμα, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς. Ξεκινώντας από αυτή την ιδέα της ενίσχυσής τους, να κάνω δύο ερωτήσεις για δύο βασικά εμπόδια που υπάρχουν σε αυτό το δρόμο, σε αυτή την πορεία ενίσχυσης και ενδυνάμωσης ε, των Αθήγκανων και γενικά των ε, διοκόμενων αυτών κοινοτήτων και απομονωμένων κοινοτήτων. Καταρχάς, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οι ίδιοι οι Ρωμά ή τα γνωρίζουν ελάχιστα. Δεν ξέρουν ποιος τους εκπροσωπεί στην κοινωνία. Και επομένως ε, έχουν τη δυνατότητα σπάνια να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν αυτά τα δικαιώματα. Κατά τη γνώμη σας, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτήν την κατάσταση. Γιατί η γνώση των δικαιωμάτων είναι το πρώτο βήμα για να αποκτήσει κανείς δύναμη. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το θέμα της συλλογή των δεδομένων. Είναι πολύ σημαντική η συλλογή, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων. Παρότι είναι προφανές ότι όλοι οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολίτες, είναι σημαντικό το πώς συλλέγονται τα δεδομένα για αυτούς. Παράλληλα, υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα και καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει πρόβλημα για τη συλλογή των δεδομένων. Το είπατε αυτό και στο ελεκτικό συνέδριο. Γιατί πάντα οι ευάλωτες κοινότητες φοβούνται ε, τις ε, απογραφές. Αυτό από την Παλιά Διαθήκη συμβαίνει έτσι. Φοβούνται τον εντοπισμό, φοβούνται τις απογραφές. Για μένα δεν έχει λυθεί αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα της συλλογής των δεδομένων. Γιατί συχνά αυτές οι κοινότητες, η κοινότητα των Ρωμά προκειμένου, έχουν την τάση να αποσιωπούν το γεγονός ότι είναι Ρωμά. Υπάρχει πρόβλημα στην κοινότητα λοιπόν, η οποία δεν αναγνωρίζεται καν. Αυτό συνέβαινε και με τους Εβραίους στην Ευρώπη. Δεν συμβαίνει πια, γιατί οι Εβραίοι πια έχουν μια πολύ, μια πολύ ισχυρή θέση στην κοινωνία, αλλά με τους Ρωμά εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα της αναγνώρισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Η κυρία Στίβενς. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Άκουσα την παρουσίαση της κατάστασης των Ρωμά στην Ανατολική Ευρώπη. Πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση των Ρωμά. Αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε το τι μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι οι Ρωμά. Αν δούμε τους ανθρώπους που έρχονται στην Δυτική Ευρώπη, συγκεκριμένα στη δική μου την πόλη, την Γάνδη, όπου έχουμε μεγάλο πληθυσμό Ρωμά, ενηλίκων και παιδιών. Ήμουν, ξέρετε, εγώ και παλιά δημοτικό σύμβουλο στην ε, πόλη μου και δεν πρέπει να υποτιμούμε τις προσπάθειες που έχει κάνει το Βέλγιο για να υποδεχτεί αυτούς τους ανθρώπους και θυμάμαι πως είχε ρωτήσει κάποτε ο Δήμαρχος ε, την ε, Κομισιόν το τι γίνεται με τα κονδύλια για τη στήριξη των Ρωμά στην Ανατολική Ευρώπη και από ό,τι φαίνεται ότι δεν χρησιμοποιούνται πλήρως τα κονδύλια από τις ε, αρχές εθνικές και τοπικές στις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Γιατί οι αρχές εκεί πέρα δεν έχουν την ικανότητα ή ίσως και τη θέληση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, για να κάνουν κάτι παραπάνω. Γιατί βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση εθνική στα ευρωπαϊκά έργα 10 με 20% ε, και Γι' αυτό το λόγο δεν ε, χρησιμοποιούνται συχνά και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εν τω μεταξύ, η πόλη της Καναδής ε, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτά τα κονδύλια. Εάν μετά από ένα-δύο γύρους μένουν ανεκμετάλλευτα στην Ανατολική Ευρώπη, γιατί να μην γίνουν με τα ίδια λεφτά έργα για τους Ρωμά στη Δυτική Ευρώπη. Ε, όπως σας είπα έχουμε αρκετούς ε, ε, Ρωμά και δεν έχουμε τα κονδύλια αυτά στην διάθεσή μας. Τα κονδύλια αυτά είναι διαθέσιμα μόνο για ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ξεχωριστός προπολογισμό, αλλά εάν μένουν τα χρήματα ανεκμετάλλευτα, γιατί να μην διατεθούν για έργα για τους Ρωμά στην ε, Δυτική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ κυρία Σουίνμπερν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε με... για την έκθεση. Λυπούμεθα που δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση για τους Ρωμά μέσα αυτά τα χρόνια. Για ένα κανεί μέλο μέλος της Ευρωπαϊκής θα πρέπει να πληρεί και να σέβεται τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Και τα τρία βασικά κριτήρια είναι η πολιτική, η οικονομική και η διοικητική πτυχή που πρέπει να σεβόμαστε. Ε, συχνά μιλάμε επίση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και λέμε ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστά παντού, αλλά βλέπουμε ότι συχνά δεν τα σεβόμαστε εμεί εδώ στα κράτη-μέλη. Η Ρουμανία εδώ και 10 χρόνια είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την αρχή κλείσαμε τα μάτια σε αυτά που συμβαίνουν στη χώρα αυτή και θεωρούσαμε ότι τελικά θα συμμορφωθεί με τα κριτήρια τη Κοπενχάγη. αλλά 10 χρόνια μετά τι συνέβη, ε, κάναμε τα πάντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε το επίδοση χρηματοδότησης για το κοινωνικό ταμείο και όμως τίποτα δεν βοήθησε. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις χώρες που δεν πληρούν τα κριτήρια. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους. Μόνο οι χώρες οι ίδιες μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες τους. Η Σουηδία, η χώρα μου, εκεί είχαμε πολλούς ε, ξένους που ήρθαν στις χώρες μας, στη χώρα μας. Καθόντουσαν ε, δεξιά και αριστερά έξω από μαγαζιά κτλ. Ε, διαβάσαμε εκθέσεις για σωματεμπορία, για λαθρεμπόριο ανθρώπων. Εκμεταλλεύονται κάποιοι τους κανονισμούς του Δουβλίνου. Έχουμε ανθρώπους ξένους οι οποίοι δεν έχουν στέγη, κάθονται έξω στο κρύο κτλ. Έχουν πέρασει πάρα πολλά χρόνια. Τι κάνουμε. Δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Η Σουηδία τι μπορεί να κάνει. Θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια στα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Σας παρακαλώ απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις. Τέλος. Η κυρία Σίπολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω την αλήθεια, έχω χάσει την ψυχραιμία μου. Δηλαδή τα άκουσα αυτά και ζήτησα το λόγο γιατί εντάξει θέλω να ρωτήσω, εντάξει, αλλά συγκεκριμένα τι έχει αλλάξει στην καθημερινότητα των ανθρώπων από το 2011 μέχρι το 2016. Και μετά ακούστηκε η απάντηση από τον εκπρόσωπο, ε, μάλλον δεν ακούστηκε η απάντηση από τους εκπροσώπους Κομισιόν. Ακόμα και το θέμα του ορίου της στόχιας από το 90% στο 80% ε, κάνατε όντως κάτι ή απλά αλλάξε ο ορισμό. Δηλαδή είναι πραγματικά τραγική αυτή η απλα αλλαξε ο ορισμος δηλαδη ειναι πραγματικα τραικη αυτη η εικονα Και αν σκεφτούμε ότι αυτά τα νούμερα αφορούν ανθρώπους και το πώς ζουν στην Ευρώπη. Και ακούμε μετά η Κομισιόν θέλει και άλλα δεδομένα. Ε, μα πόσα δεδομένα χρειαζόμαστε για να αναγνωρίσουμε ότι η ζωή πολλών ανθρώπων στην Ευρώπη είναι αφόρητη. Ε, δεν χρειάζεται καμία διάσκεψη και άλλα στατιστικά στοιχεία. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα λάβουμε μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Άλλη μία διάσκεψη και άλλα δεδομένα δεν θα μας βοηθήσουν. Και μία τελευταία παρατήρηση. Όλοι έχουμε διαδίκτυο. Κοίταξα, μιλάμε για χριστιανισμό και τα Ματθαίος 25 ε, και τα λοιπά, τα ξέρετε. Αγαπάτε τον πλησίον ε, ως εαυτόν. Ε, αν πάρουμε αυτό ως μέτρο, δεν είμαστε χριστιανική Ήπειρος. Εδώ πέρα παραβιάζεται κατάφορα η αξιοπρέπεια των ανθρώπων και κάνουμε τη μία διάσκεψη μετά την άλλη. Εγώ δεν θέλω άλλη μία έκθεση και άλλη μία διάσκεψη. Πρέπει επιτέλους Κομισιόν και κράτη-μέλη να μιλήσουν με ποια συγκεκριμένα μικρά έργα θα βοηθήσουν τους ανθρώπους. Uh, Καλός και ωραίο τρόπος για να ολοκληρωθούν έτσι οι παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητέ. Ε, πιεζόμαστε από το χρόνο. Έχουμε 5-6 λεπτά. Ε, ξέρω βεβαίω ότι θα θέλατε να απαντήσετε έτσι πιο διεξοδικά, αλλά πιεζόμαστε. Ξεκινάμε με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη, γιατί δεν θα μπορέσω να καλύψω τα πάντα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Καταρχάς, να ξεκινήσω από το νομοθετικό πλαίσιο. Ε, από τα στοιχεία που έχουμε σύν το χρόνο, ε, όχι μόνο για την ένταξη των Ρωμά, αλλά και τις έρευνες που κάναμε για τους μετανάστες, για τους ΛΟΑΔΑ, ακόμα και για τη βία κατά των γυναικών, προκύπτει ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένα χάσμα, υπάρχει πρόβλημα με την αφύπνιση, με τη γνώση για την ομοθεσία, ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις ε, φιλετικές ισότητες υπάρχει ένα θέμα δυναμικού ε, των φορέων ισότητας για να υποστηρίξουν τα άτομα αυτά. Ούτως ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν και να καταγγείλουν περιπτώσεις μοιήσεις μεταχείρισης. Υπάρχει ένα θέμα με την εφαρμογή επίσης, ό,τι αφορά και την οδηγία για την ε, φιλετική ισότητα και την ισότητα στην εργασία. Ε, μιλήσατε για το θέμα της, του έντονου, της έντονης περιθωριοποίησης. Καλύπτουμε το θέμα αυτό στην έρευνα. Βεβαίως θέλουμε να καλύψουμε κυρίως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, όσο πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται, ε, για αυτούς τους 6 εκατομμύρια Ρωμά που ζουν στην Ευρώπη. Η αναγνώριση, όπως είπατε, ε, απαράδεκτων διακρίσεων, ε, το ιστορικό υπόβαθρο είναι και πολιτικό θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που ρίχνουν άπλετο φως στη μεταχείριση των Ρωμά ε, σε όλα αυτά τα κράτη-μέλη παλαιότερα και σήμερα. Υπάρχει θέμα εδώ πολιτική πρωτοβουλία, ούτω ώστε να υπάρξει αναγνώριση αυτού του προβλήματο. Πέρα όμω από αυτή την πολιτική πρωτοβουλία, ε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται μόνο μια δήλωση, αλλά και καθοδήγηση για την κοινωνία, για να καταλάβει έτσι όπως για να καταλάβει ας πούμε, τι βλέπει όταν βλέπει τα παιδιά ας που, πλέβουν, που παίζουν στην ε, λάσπη, ε, που κλέβουν για να ζήσουν, που ζουν στους καταβλισμούς κτλ. Ε, τα διαφορετικά ταμεία τα αναφέρατε πολλές φορές. Η εκ των προτέρων ε, αιρεσιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη. και αυτό έχει να κάνει με το πώς οι διαχειριστικές αρχές τελικά χρησιμοποιούν τη διατύπωση για να όταν ε, ετοιμάζουν ε, τις, ε, τους διαγωνισμούς, όταν το πώς ανταποκρίνονται οι τοπικές αρχές σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις διαχειριστικές αρχές και από ό,τι ξέρω η Κομισιόν ήδη κάνει μια προσπάθεια και ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια να φέρει αποτελέσματα. Να κλείσω χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες με δύο πράγματα. Σοβαρές προσπάθειες για την ένταξη των Ρωμά ξεκίνησαν πριν από 15 χρόνια, έτσι χοντρικά, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 15 χρόνια πριν. Είναι λιγότερο από μια γενιά αυτό, έτσι. Πολύ λιγότερο από μια γενιά. Και παρότι μπορείτε να έχετε την αίσθηση ότι εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι ε, αισθανόμαστε αγανακτισμένοι όταν βλέπουμε ανθρώπου να ζουν εδώ στην Ευρώπη σε συνθήκε τρίτου κόσμου. Σκεφτείτε πόσο χρόνο χρειάζεται ούτω ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους ε, να βγουν από την κατάσταση, να ενισχυθούν, όχι να του δώσουμε λιμοσύνη ας πούμε, να του βγάλουμε, να τους δώσουμε τα στοιχεία, τα εργαλεία για να βγουν από αυτήν την κατάσταση φτώχεια. Αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα στοιχεία και χρειαζόμαστε βέβαια περισσότερη πρόοδο. Κλείνοντα. κλείνω με δύο πράγματα που νομίζω ότι είναι στον πυρήνα τη προσπάθεια ένταξη των Ρωμά. Το ένα είναι η αξιοπρέπεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η βασική δουλειά για την ένταξή του θα πρέπει να εδράζεται στην αξιοπρέπεια και, το... και να είμαστε σίγουροι ότι υποστηρίξουμε αυτή την αξιοπρέπεια ε, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε την ενίσχυση και την ένταξη να τα βάλουμε μαζί. Τα έχουμε πει πολλές φορές, ο κόσμος έχει βαρεθεί να τα ακούει, αλλά πραγματικά πρέπει να εστιάσουμε στην εμπιστοσύνη. Ε, αυτή τη στιγμή πολλές κοινότητες Αθήκανων δεν ε, εμπιστεύονται τους πολιτικούς, ακόμα και όταν κάνουν προσπάθεια για να τους ε, εντάξουν μέσα από προγράμματα, μέσα από project, ε, μέσα από έργα. Πρέπει να κάνουν προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο. Και επίσης δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη μεταξύ των τοπικών αρχών ότι οι επενδύσεις που θα κάνουν θα έχουν ένα βιώσιμο αποτέλεσμα. Και καλό αποτέλεσμα βέβαια. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί δημιουργούν μια πολύ ζωφερή εικόνα, αλλά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και όπως είπα, η ένταξη, το θέμα, το θέμα της ανάπτυξης, το θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, όλα αυτά για να φέρουν αποτελέσματα, για να τα προωθήσουμε και να φέρουν αποτελέσματα πρέπει ε, να δεχτούμε ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Κύριος Σμιτ, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με την παρατήρηση της κυρίας Σπινέλη. Ανέφερε το ότι ε, πολλοί Ρωμά κρύβουν την ταυτότητά τους. Εκεί πέρα είναι το πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι στην Ευρώπη δεν μπορούν να είναι περήφανοι για την ε, καταγωγή τους, τότε έχουμε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο δεν υπάρχει εδώ και 10, 15, 20 χρόνια. Ε, υπάρχει κυριολεκτικά εδώ και αιώνες οι προκαταλήψεις αυτές και αυτές πρέπει να καταπολεμήσουμε. Κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να κάνει η Κομισιόν εδώ πέρα από τις Βρυξέλλες σε κάθε χωριό της Ευρώπης όπου υπάρχει αυτή η δυσπιστία. Πρέπει αυτό το πράγμα να συμβεί μέσα στα μυαλά των ανθρώπων και έρχομαι άρα στα συγκεκριμένα ερωτήματα που ακούστηκαν. Ρωτήσατε, κύριε Πρόεδρε, αν επαρκεί το νομικό πλαίσιο, το οποίο υπάρχει ήδη εδώ και κάποια χρόνια η οδηγία για τη φιλετική ισότητα, αλλά και η απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου. Θεωρώ πως ε, το ερώτημα πρώτα απ' όλα πρέπει να τεθεί διαφορετικά. Τα μέσα αυτά εφαρμόζονται πρώτα απ' όλα. Στα κρατημέλη και απάντηση είναι μάλλον όχι και θεωρώ πως εδώ είναι πολύ σημαντικό τα μέσα τα οποία έχουμε σήμερα και τα οποία από το 2014 έχουν μεταφερθεί πλήρως στο νομικό πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να χρησιμοποιηθούν όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Και κάτι το οποίο ανέφεραν αρκετοί βουλευτές. Οπωσδήποτε υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα σε κράτη-μέλη και μάλιστα όχι μόνο όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και όσον αφορά και την εφαρμογή του δικαίου. Αυτό το οποίο ε, δεν βλέπουμε όμως είναι ότι είναι ε, κάτι το οποίο γίνεται εσκεμένα. Είναι περισσότερο μια αδράνεια και μια αδιαφορία των αρχών που δεν λαμβάνουν τα σωστά μέτρα έτσι ώστε οι νόμοι παραδείγματος χάρη για την προστασία κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων να εφαρμοστούν. Αλλά αυτά τα οποία λέτε, ε, ε, καταναγκαστική στήρωση, μα για το όνομα του Θεού δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά γίνονταν στην κομμουνιστική δικτατορία. Αν υπήρχε τέτοιο πράγμα σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ε, υπάρχουν όμως άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Αναφέρατε πράγματι χωριστά σχολεία. ίσως ε, όχι από πρόθεση, αλλά υπάρχει μια κατάσταση η οποία ε, περιγράφεται ως ε, διαχωρισμός στα σχολεία. Και τους λέμε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό ως ε, κομισιόν, το έχουμε τονίσει στα κράτη-μέλη και μπορώ να σας πω ότι κανένα από τα κράτη-μέλη δεν επιμένει ότι είναι σωστή αυτή η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα βρούμε τα σωστά μέτρα για να τερματιστεί ε, αυτός ο διαχωρισμός ο οποίος υπάρχει. Και βεβαίως το ίδιο ισχύει και με την πρόσβαση στα έγγραφα ταυτότητα. Συμφωνώ είναι αναξιοπρεπές σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς δελτίο ταυτότητας. Κάτι άλλο ε, σημαντικό που ανέφεραν αρκετοί βουλευτές ε, αυτή η ενδυνάμωση που λέτε να τους βοηθήσουμε να βοηθηθούν από μόνοι τους. Ε, προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε Παραδείγματο χάρη υπάρχει τώρα ένα κοινό πρόγραμμα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, λέγεται Youthstrom, όπου έχουμε στόχο ειδικά οι γυναίκες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, οι γυναίκες Ρωμά και να ενδυναμωθούν έτσι. Και εδώ πέρα ακριβώς ε, βασιζόμαστε στην υφιστάμενη νομοθεσία. Ξέρετε πως ε, έχουμε και τους φορείς της ισότητας ε, που είναι υποχρεωμένοι με βάση την οδηγία κατά του ρατσμού να κινητοποιηθούν στο θέμα αυτό και νομίζω πως αυτά είναι αυτά τα οποία μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενοι νόμοι θα εφαρμόζονται Κάτι από το οποίο απέχουμε ακόμα πολύ όσον αφορά τους ε, Ρώμα. Ε, τώρα η αλλαγή της νοοτροπίας θα πρέπει να γίνει στην κάθε χώρα. Όσον αφορά τώρα την δομή, υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που συμφώνησε Συμβούλιο με Κοινοβούλιο και ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί για την ε, αναδιανομή των κονδυλίων για αυτό που ρωτήσατε. Οπότε δεν θέλω να δημιουργηθεί εντύπωση ότι κάποιος ε, κάνει τα στραβά μάτια εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια να ασχολούμαστε σοβαρά με αυτό το θέμα. Το 2011 υπάρχει η στρατηγική και πρέπει να συνεχίσουμε και τα, τα μικρά βήματα προς σωστή κατεύθυνση πρέπει να τα αναφέρουμε και να εφαρμοστεί αυτή η στατική. Σας ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ και τους δύο καλεσμένους μας. Έχουμε και ένα επιπλά στην σε διάταξη, αυτό που έθεσε ο κύριος Άλμπρεχτ. Ε, και ζήτησαν και δύο συνάδελφοι το λόγο. Καθυστερούμε τον κύριο Τεμπρέ. Παρακαλώ, πολύ σύντομα. Ναι, δεν συμφωνώ με τη δήλωση ότι κανείς και μένα δεν επιδεινώνει αυτή την κατάσταση. Απλώς τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα, δεν αναλαμβάνουν δράσεις. Λυπάμαι, αλλά είναι θέμα βούληση των κρατών μελών το ότι δεν κάνουν κάτι μερικέ φορέ, ότι δεν κάνουν τίποτα. Και άρα είμαστε υπεύθυνοι για αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Και αν μιλάτε για ένα γενικό κανόνα και μία υποχρέωση να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, ενώ έχουμε παιδιά που μένουν σε απομακρυσμένα χωριά, πολύ μακριά από το σχολείο, δεν υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες, δεν υπάρχουν δημοτικές συγκοινωνίες, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αυτοκίνητο, τότε μην μας λέτε ότι «Α, οι καημένοι δεν παίρνουν σωστή κατεύθυνση». Υπάρχει απροθυμία των κρατών μελών θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην βρίσκουμε προσχήματα για να παραμένουμε στα ίδια. Η Σωράγια παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την uh, Σίπελ. Γι' αυτό, αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά, σε ολόκληρη την κοινωνία. Θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλα τα μέλη της κοινωνίας και να έχουμε πιο συντονισμένες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε αυτή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλου. Θα θέλαμε μια ομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συντονίζει τις εργασίες των επιμέρους γενικών διευθύνσεων. Γιατί να αλληλένδεται αυτά τα θέματα. Δεν έχει νόημα να να μιλούμε για την εκπαίδευση αγνώντας τους, τις συνθήκες διαβίωσης ή τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία. Μιλήσαμε για τριτοκοσμικές συνθήκες διαβίωσης στην καρδιά της Ευρώπης. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Και παρόμοια προβλήματα έχουμε και στη Σουηδία, όπως και στη Γαλλία και τη Βουλγαρία. Παντού τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να νιώθουν περήφανοι για την ιστορία τους, για την καταγωγή τους και θα πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη από τους ανθρώπους ε, που καταπατήσαμε τα δικαιώματά τους για τόσα χρόνια. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν αναλάβουμε τις ευθύνες μας, θα συνεχίζουμε να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων διακρίσεων και ρατσισμού ή ρατσιστικής ρητορικής. Γιατί Πολλοί δεν τρέπονται να μιλούν κατά των συμπατριωτών τους. Θα πρέπει τέτοιου είδους φαινόμενα να τα καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ Σωράγια. Ξέρω ότι ζήτησες και εσύ το λόγο Μπάρμπαρα, αλλά αν δώσω το λόγο σε όλους που το ζήτησαν, θα μετανιώσετε που με επανεκλέξατε. Άντε, εν πάση περιπτώσει, μία πρόταση μόνο μας, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι θα με μισήσεις τώρα, αλλά να πω κι εγώ μία πρόταση. Τελικά έχω το δικαίωμα ή όχι. Όχι, πρέπει να τελειώσουμε. Θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω. Γνωρίζω ότι θα θέλατε κι εσείς να απαντήσετε στα τελευταία σχόλια. Το φαντάζομαι, αλλά... Α, μείνετε στο πνεύμα των σχόλιων αυτών. Έχουμε ευρωβουλευτές από κράτη-μέλη που έχουν ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και έχουν πλούσια πείρα, γιατί είναι πολύ εξοικειωμένοι με το θέμα, το ίδιο με εσά. Και ήταν χρήσιμη αυτή η ενημέρωση, γιατί πραγματικά είναι πολύ κακή η κατάσταση. Δεν υπάρχει εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων από τα κράτη-μέλη. Και μάλιστα μερικές φορές έχουμε και επιδείνωση σε σχέση ε, με τα προηγούμενα στοιχεία, ιδιαίτερα στο θέμα της φτώχειας. Το θέμα της φτώχειας έχει επιδεινωθεί για την κοινότητα των Ρωμά. Οπότε η κατάσταση είναι πολύ κακή, η εφαρμογή δυστυχώς ε, μένει πίσω, οπότε ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς. Πάντως, αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι θα ξαναφέρουμε το θέμα ε, πολύ σύντομα στην ημερήσια διάταξη. Δεν θα το αφήσουμε κατά μέρους. Σας ευχαριστώ για την ε, προθυμία σας και θα σας ε, ξανακαλέσουμε στο εγγύς μέλλον για να δώσουμε συνέχεια. Και σας ευχαριστώ όλους για τις ε, πολύ ε, έντονες παρατηρήσεις και το ζωηρό ενδιαφέρον. Περνάμε στο επόμενο θέμα, σε αυτό που προσθέσαμε και που εγκρίναμε να προσθέσουμε. Να δώσουμε δηλαδή ένα πεντάλεπτο, πέντε-έξι λεπτά στους δύο δικηγόρους που παρακολουθούν την κατάσταση του κυρίου Έντουαρτ Σνόουδεν. Θα μας ενημερώσει, γιατί έχουμε και το ψήφισμα της 12 η Μαρτίου για το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα την έκθεση πρωτοβουλίας για τις μαζικές παρακολουθήσεις. Ξέρω ότι το θέμα αυτό ενδιαφέρει πολλούς και το ακροτηριό μας ε, από το διαδίκτυο. Ένα πεντάλεπτο παρακαλώ, συνοπτικά, πείτε μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Μπεν Βάιζον από την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών και έχουμε τον συνάδελφο από το Συνταγματικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαστε νομικοί σύμβουλοι του Έντουαρτ Σλαούδεν και τον ε, εκπροσωπούμε στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, σας μεταφέρω του θερμού χαιρετισμού του Έντουάρτ Snowden που εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για το ψήφισμά σα του 2015 που τον αναγνώρισε ως ε, Διεθνή Εκτεπιστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ευθύνεται έκκληση στα κράτη-μέλη να του χορηγήσουν προστασία και παρόλο που υπάρχουν αρκετέ διαφωνίε ε, στι κοινωνίε μα για το τι είδου παρακολούθηση, πολιτικέ παρακολούθηση θα πρέπει να εφαρμόζουν οι χώρε. υπάρχει η ευρεία συμφωνία ότι στι ελεύθερε κοινωνίε τέτοιου είδου αποφάσει θα πρέπει να γίνονται μετά από ανοιχτή δημόσια συζήτηση και όχι και κλεισμένο το θηρόν από οι μυστικέ υπηρεσίε που λαμβάνουν τι αποφάσει παρασκηνιακά και πίσω από την πλάτη μα. Είχαμε ελπίσει πριν ε, το τέλος της θητείας ε, του Πρόεδρου Ομπάμα να δοθεί μια δίκαιη λύση στην υπόθεση Snowden στις ΗΠΑ. Δυστυχώς δεν συνέβη κάτι τέτοιο και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ε, σοβαρές απειλές με βάση τον ε, νόμο για την κατασκοπή από το πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για, για πώληση μυστικών σε ξένες δυνάμεις. Τώρα έχουμε ένα νέο πρόεδρο που ανα, ανήκει ήδη στο Twitter ότι θα πρέπει να εκτελεστεί ο κύριος Σνόουντεν και μάλιστα ε, όρισε ως διευθυντή της CIA κάποιον που συμμερίζεται αυτή την άποψη. Θα πρέπει να εκτελεστεί για τις πράξεις του κ. Σνόουντεν. Εμείς βρισκόμαστε εδώ ελπίζοντας ε, ότι δεν θα ξεχάσετε τον ε, Έντουαρτ Σνόουντεν, γιατί έχει πολλά να συμβάλλει, να συνεισφέρει. Θα ήθελε πολύ να είναι εδώ αυτοπροσώπος ο ίδιος και ελπίζει να έχει την ευκαιρία αυτή σύντομα στο σχετικά εγγύς μέλλον. Έχει πλούσια εμπειρία που μπορεί να σας την παρουσιάσει, ώστε να μπορέσετε να ασχοληθείτε με το περίπλοκο θέμα της μαζικής παρακολούθησης της ελεύθερης κοινωνίας. Και ευελπιστώ ότι η Επιτροπή σας θα στηρίξει αυτό το ψήφισμα και θα εντείνει τις εκκλήσεις προς τα κράτη-μέλη να χορηγήσουν προστασία στον κύριο Σνόντεν. Ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσετε. Όπως είδατε δεν εξατλήσαμε καν το εξάλεπτο. Σας ευχαριστώ και καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση του θέματος. Ξέρω ότι σας περιμένουν και άλλες συναντήσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς θα προχωρήσουμε στα δικά μας θέματα. Και ο κύριος Άλμπρεχτ και άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να σας μιλήσουν έχουν την ευκαιρία να το κάνουν γιατί έχετε διάφορες επαφές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε μπορείτε να έχετε σε επικοινωνία με το γραφείο του κυρίου Άλμπρεχτ για να δώσετε και την σύντομη παρουσίαση που κάνατε. Περνάμε τώρα στο σημείο 10, τις ε, ερωτήσεις που ζητούν γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για ερωτήσεις του κυρίου Ντεπρέ για την συμπερίληψη των στοιχείων στο σύστημα ΣΥΣ και στη Eurodac για αποφάσεις επιστροφών. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας κύριε Ντεπρέ. Εδώ Έχουμε λάβει τις απαντήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 13 Ιανουαρίου. Βέβαια, η διορία για τις ερωτήσεις αυτές είχε εκπνεύσει όσα είστε. Θέτουμε εμείς τα ζητήματα, μια και έχει λήξει προθεσμία για να το κάνουν τα κρατη Ο Ζεράρ Πρέ για να μας κάνει μια ενημέρωση και παρουσίαση της ερώτησής του. Ευχαριστώ. Ε, είμαι σε δύσκολη θέση γιατί είναι η δεύτερη-τρίτη ή φορά που εκπρόθεσμα μας απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως γιατί θέλουν συνέχεια να ακούν τη δικιά μου φωνή στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών γιατί θα μπορούσε καλή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει στείλει γραπτός ε, την απάντησή της εμπρόθεσμα μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, πιο σοβαρά τώρα. Θα ήθελα να σας κάνω μια παρουσίαση για να παρακολουθήσουν το θέμα οι συνάδελφοι. Λέω λοιπόν ότι το άρθρο 14 της ε, πρότασης για τη Eurodac προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να ε, ε, λάβουν βιομετρικά στοιχεία όλων των υπηκών των τρίτων χωρών που παράτυπα διαμένουν στην επικράτειά τους. Παράλληλα, το άρθρο 6 της Οδηγίας για τις Επιστροφές προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνουν απόφαση επιστροφής ε, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν παράτυπα στην επικράτειά τους. Όσοι λοιπόν διαμένουν παράτυπα ε, στα κρατημέλη, ε, εμπίπτουν ταυτόχρονα και στο Eurodac και στο σύστημα SIS, γιατί ε, προβλέπεται ότι στο νέο SIS θα περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις περί επιστροφής. Τι προσθέτει λοιπόν αυτή η διπλή καταχώρηση και στη Eurodac και στο σύστημα SIS. Υπάρχουν κάποιοι που θα πρέπει να είναι στο Eurodac δυνάμει του άρθρου 14 αλλά που δεν ε, αποτελούν το αντικείμενο απόφαση επιστροφής και άρα δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στο ΣΥΣ. Και αν, ε, αν υπάρχουν άνθρωποι που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, τότε τι προσθέτει αυτή η διπλή καταχώρηση και η καταχώρησή του στο Eurodac. Δηλαδή έχουμε δύο συστήματα που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία. Έχω λάβει την ε, απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επειδή έχω και συμπληρωματική ερώτηση, ήθελα να μας την παρουσιάσει πρώτα αυτή την απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Déjà vu, έχω την αίσθηση ότι κάπου τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Ο κύριος Κοέλιο. Θα προτιμούσα να θέσω την συμπληρωματική μου ερώτηση αφού ακούσω την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλώς. ο εκπρόσωπο τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων που θα απαντήσει την ερώτηση του κ. Ντεπρέ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σα. Μαόρο Γκαλιάρντι ονομάζομαι. Εγώ θα απαντήσω τελικά στην ερώτηση του κ. Ντεπρέ από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την ε, απάντηση σε αυτή την κοινοβουλευτική ερώτηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντεπρέ για την ερώτησή του, που είναι πολύ εύστοχη και επίκαιρη για τη συζήτηση που γίνεται για τη Eurodac και το ΣΥΣ. Όπως αναφέρεται και στο επεξηγητικό σημείωμα που συνοδεύει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος της Eurodac είναι να διευκολύνει την ταυτοποίηση ε, και τα στοιχεία για τους παράτυπους ε, μετανάστες ε, εν ώψη της πιθανής επιστροφής τους. Και κυρίως όσους χρησιμοποιούν πλαστά στοιχεία για να αποφύγουν τη χορήγηση των σωστών στοιχείων και κινούνται, διακινούνται παράτυπα μεταξύ των κρατών μέλων. Με την πρόταση αυτή θα μειώσουμε τη διαδικασία των επιστροφών και την περίοδο κράτησης αυτών των μεταναστών, των παράτυπων μεταναστών και θα καταπολεμήσουμε με τα βιομετρικά στοιχεία απάτες ε, περί ταυτότητα. Τώρα, η πρόταση για την ε, για τις προειδοποίησεις ε, για τις προτάσεις επιστροφής στο σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν, το ΣΥΣ δηλαδή, που υποβάλαμε πριν από λίγε εβδομάδε, ο στόχο είναι διαφορετικό. Είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτέ τι αποφάσει επιστροφή. Και να δούμε ότι πραγματικά έχει υλοποιηθεί αυτή η απόφαση τη επιστροφή. Πέραν των προειδοποίησεων λοιπόν αυτών, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να ε, κοινοποιούν και επιπλέον στοιχεία για τις επιμέρους υποθέσεις μέσω του ε, των γραφείων τους, ε, επιτρέπονται στις εθνικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με βάση την οδηγία περί επιστροφών και τα στοιχεία της Eurodac. Επίσης θα διευκολύνουν την εφαρμογή των κανόνων για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων επιστροφής. Οπότε τα στοιχεία για τον ίδιο παράτυπο μετανάστη θα υπάρχουν και στη Eurodac και στο σύστημα πληροφοριών του Schengen, το SIS. Βέβαια, και εδώ είναι η σημαντική διαφορά, θα είναι προσιτό το σύστημα μόνο σε διαφορετικές αρχές για διαφορετικούς στόχους αυτά τα δύο συστήματα και θα είναι διαφορετικές και οι ε, διορίες κράτησης αυτών των στοιχείων και φύλαξη αυτών των στοιχείων και αυτό γίνεται με στόχο την, τον περιορισμό σε ό,τι αφορά τη χρήση ε, και την συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων. Οπότε τα δύο αυτά ε, εργαλεία είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και δεν αλληλοεπικαλύπτονται. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τις προειδοποίησεις, για τις επιστροφές, αυτά θα μπουν στο ΣΥΣ μετά την έκδοση της απόφασης περί επιστροφής. Ενώ τα στοιχεία στη Eurodac μπορούν να καταχωρηθούν και σε πρώτερη φάση, άσχετα με την πιθανή απόφαση επιστροφής. Οπότε, αν ένας παράτυπος μετανάστης ε, ε, ε παρόλο που μια απόφαση για το ΣΥΣ δεν, δεν θα υπάρχει γιατί δεν θα έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, θα υπάρχουν τα στοιχεία του στη Eurodac. Οπότε, ε, άλλη περίπτωση θα είναι μια απόφαση ε, επιστροφής να, αποφα... να αφορά της χώρας για ένα ποινικό αδίκτυμα, οπότε σε τέτοια περίπτωση θα περιλαμβάνεται η απόφαση στο ΣΥΣ, αλλά θα περιλαμβάνεται και στη Eurodac. Ελπίζω να διευκρινίστηκε η απάντηση προς τον κύριο Ντεπρέ. Πριν επανέλθω στον κύριο Ντεμπρέ, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κοέλιο για τη συμπληρωματική ερώτηση. Έχετε ερώτηση, κύριε Κοέλιο. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεπρέ. <clears throat> Πρόεδρε, συνήθω ε, συμφωνώ με τον Ζεγάρ Ντεπρέ. Αλλά όχι σήμερα. Καταλαβαίνω την απάντηση που έδωσε η Κομισιόν. Ο στόχος των δύο εργαλείων, των δύο κειμένων, είναι διαφορετικό. Το ΣΥΣ και το Eurodac. Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία για επικάλυψη διαδικασιών, τότε καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στο σύστημα πληροφοριών του ΣΕΝΚΕΝ, στο ΣΥΣ. Ε, γιατί είναι πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο ευρύ ως προς τους στόχους σε σχέση με το Eurodac. Αν θέλουμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, δεν συμφωνώ με την άποψη κύριε Ντεπρέ, αλλά αν θέλουμε να αποφύγουμε τι επικαλύψει, θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν, το ΣΥΣ, και όχι το αντίθετο. Έχουμε την ευκαιρία, ή μάλλον θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε πολιτικέ αποφάσει και νομοθετικέ αποφάσει όταν αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για το ε, ΣΥΣ 2. Η πρόταση είναι στο τραπέζι, έχει κάνει την πρόταση της η Κομισιόν και μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τότε στο πλαίσιο της Επιτροπής μας και να πάρουμε την απόφαση για την ε, αρχιτεκτονική και τη δομή που θέλουμε να φτιάξουμε για το ΣΥΣ και το Eurodac, ούτως ώστε να απαντήσουμε μεγάλη αποτελεσματικότητα ε, σε, αυτές, σε αυτά τα θέματα αποφάσεων επιστροφών. Ο Ζεγάρ. Μπορείς να απαντήσεις και στον ερώτηση του κυρίου Κοέγιο, παρακαλώ. Πρόεδρε, λυπάμαι που ο Κάρλος δεν συμφωνεί <laughs> αυτή τη φορά μαζί μου. Ε, εγώ δεν διαφωνώ μαζί του όμως. Ε, αν θέλουμε να επικεντρωθούμε κάπου, όντως θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ΣΥΣ. Μία παρατήρηση και δύο έχω να κάνω. Καταρχάς, διαπιστώνω ότι η τροποποίηση του σύστηματος Eurodac σημαίνει ότι για κάθε άτομο που βρίσκεται σε παράνομη ε, διαμονή, 10 ε, δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου θα βάλουμε τέσσερα δακτυλικά αποτυπώματα και ένα του προσώπου. Γιατί αυτό έχει επίπτωση στο σύστημα του, στη λειτουργία του συστήματος. Ποιος είναι ο λόγος. Η Κομισιόν προσπαθεί να ενοπίσει όλα τα συστήματα. Ε, δύο, σε σχέση με την απάντηση. Εάν διαβάσω τις κατηγορίες προσώπων που θα, μπορούσαν να, που θα μπορούσε να αφορά αυτό το θέμα. Κομισιόν. Έχετε μια ιδέα για την αξιολόγηση του αριθμού των ατόμων που θα μπουν στο ΣΥΣ και όχι στο Eurodac. Έχετε μια ιδέα για τα άτομα, τον αριθμό των ατόμων που θα είναι στο Eurodac και, όχι στο ΣΥΣ. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα υπάρχουν και τόσα πολλά. Η τροποποίηση όμως του συστήματος Eurodac θα ε, κοστίσει 29 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η επικάλυψη λοιπόν είναι απαραίτητη. Επιμένω στο ερώτημά μου. Χρειάζεται. Ευχαριστώ, Ζεράρ. Κομισιόν. Μπορείτε να απαντήσετε. Σε αυτά τα επιπρόσθετα ερωτήματα του κυρίου Ντεπρέ. Αλλά σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ για Κομισιόν να απαντήσω καταρχάς στο δεύτερο ερώτημα. Ο λόγος είναι ο ίδιος. Εμείς θεωρούμε ως Κομισιόν ότι, ότι έχει προσθέμενη αξία το να έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις τις πληροφορίες και στα δύο συστήματα, λόγω των διαφορετικών σκοπών που εξυπηρετούν οι δύο βάσεις δεδομένων, το ΣΥΣ και το Eurodac. Η ιδέα πίσω από το ΣΥΣ και την πρόταση του ΣΥΣ, το να βάλουμε νέες καταχωρήσεις ε, επιστροφών δεν είναι μόνο να έχουμε πληροφορία, πληροφορίες για το συγκεκριμένο άτομο, το ώστε να μπορούμε να το ταυτοποιούμε, αλλά να βοηθήσουμε τις ε, διοκτικές αρχές και να βοηθήσουμε να εφαρμοστεί η απόφαση επιστροφής. Και τελικά να λάβουμε τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα, ούτω ώστε να απομακρυνθεί το άτομο. Και να κλείσουμε το φάκελο επιβεβαιώνοντας την έξοδο του ατόμου από την περιοχή Σέγγεν, δηλαδή να επιβεβαιώσουμε ότι πέρασε από ε, σημείο στα εξωτερικά ε, σύνορα. Ενώ στο Eurodac είμαστε σε τελείως διαφορετικό πλανήτη. Θέλουμε να ταυτοποιήσουμε και να δώσουμε ε, στοιχεία και δελτία, ας πούμε, συγγνώμη, ταυτότητα σε ένα άτομο το οποίο προσπαθεί να πει ψέματα για την ταυτότητά του. Σε σχέση με την, δεύτερη, με την πρώτη συμπληρωματική ερώτηση, ναι, σημειώνω ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις προτάσεις. Και σας υπενθυμίζω ότι γίνεται ακόμα δουλειά ε, στο επίπεδο, στην ομάδα υψηλού επίπεδου για την διαλειτουργικότητα. Εμείς παρακολουθούμε τη δουλειά της ομάδας υψηλού επίπεδου και θα συνεχίσει να εργάζεται αυτή η ομάδα ε, μέσα στο 17. Ζεγάρ, θες να επανέλθεις? Θα επανέλθω, Πρόεδρε, στο μέλλον και για τον αριθμό των δαχτυλικών αποτυπωμάτων και θα σχολιάσω και την απάντηση που μου δόθηκε. Ως ο νουπο. Θα ετοιμάσω και επιχειρήματα για το θέμα αυτό. Thank you very much. Ευχαριστώ. Και, κύριε, και σας κύριε Κοέγιο. Είσαστε και δύο πολύ έμπειρα μέλη. Έχω την αίσθηση κι εγώ ότι πολύ σωστά θέσατε αυτό το ερώτημα, ούτως ώστε να αξιολογήσουμε το, το του προβλήματος αυτού. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μια επαναξιολόγηση του θέματος. Ήταν χρήσιμη λοιπόν αυτή η συζήτηση, παρότι υπήρχαν ε, κάποιες διαφωνίες. Άξιζε τον κόπο η υποβολή, το να υποβληθεί αυτό το ερώτημα. Και ευχαριστώ και την Κομισιόν βεβαίως που που έδωσε απάντηση να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, δύο λεπτά. Έχω και μια δεύτερη ερώτηση εγώ. Σοβαρά. Α, συγγνώμη πρόεδρε, έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Ναι, σωστό, σωστό Ζερά, Το ξέχασα. Έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα για το ΣΥΣ. Το άρθρο 24 του κανονισμού 1987 του 2006 μιλάει για τις συνθήκες υπό τις οποίες μια καταχώρηση λόγω απαγόρησης εισόδου ή άρνησης εισόδου μπορεί να εισαχθεί από ένα κράτος μέλος στο ΣΥΣ 2. Αυτές οι προϋποθέσεις ε, είναι ευρείες. Γι' αυτό ακριβώς ε, στην αιτιολογική σκέψη, υπάρχει μια αιτιολογική σκέψη που λέει ότι θα πρέπει να εξακολουθούμε να ε, προσπαθούμε για μία εναρμόνιση ε, των διατάξεων ε, σε σχέση με τους ε, λόγους που δικαιολογούν την εισαγωγή. Γιατί αυτή τη στιγμή το κάθε κράτος είναι ελεύθερο. Το άρθρο, ένα άλλο, άρθρο τώρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, το άρθρο, άρθρο 24.5 λέει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να επανεξετάσει τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού τις διατάξεις του άρθρου 24 και βάσει τη επανεξέταση να κάνει προτάσει, τι προτάσει απαραίτητε, τι απαραίτητε προτάσει, ούτω ώστε να φτάσουμε σε ένα υψηλότερο βαθμό εναρμόνιση των κριτηρίων καταχώρηση. Το ερώτημα μου είναι απλό. Η Κομισιόν έκανε αυτή την επανεξέταση που προβλέπει το άρθρο 24 σημείο 5 και αν ναι, πότε σκοπεύει να κάνει προτάσεις για την εναρμόνιση ή για την τροποποίηση. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, Ζωά, δεν είχα δει ότι είχε και μια ερώτηση για το άρθρο 24. Κομισιόν. Έχετε κάνει την επανεξέταση αυτή του άρθρου 24. Μπορείτε να απαντήσετε στη δεύτερη ερώτηση του κ. Ντεπχέ, παρακαλώ. Yes, Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Βέλη τη λέγομαι και θα απαντήσω εξ ονόματος της ε, Κομισιόν. Δυστυχώς πρέπει να ομολογήσω ότι πράγματι δεν λάβατε την απάντηση αλλά μπορώ να δώσω κάποια στοιχεία καθώς ε, η έκθεση αξιολόγησης για το άρθρο 24 έχει ήδη δημοσιευτεί στις 25 Δεκεμβρίου και περιέχει και αυτό το σημείο αξιολόγησης του άρθρου 24 και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τα αποτέλεσματα υπάρχουν και στις ε, προτάσεις, ε, στην αναθεώρηση του μηχανισμού SIS ε, για την χρήση του για μεθοριακούς ελέγχους και για επιστροφές. Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος τελειώνει, Ζεράρα, μπορείτε να απαντήσετε. Ναι, ναι, ωραία, σας ευχαριστώ για αυτές τις πληροφορίες. Ζεράρ. Όπως είπα λοιπόν, είναι πολύ χρήσιμη συζήτηση και ευχαριστώ και πάλι την ε, Κομισιόν. Ωραία, συνάδελφοι. Κάνουμε ένα διάλειμμα ολίγων λεπτών και μετά περνάμε στο σημείο 12 με την Επίτροπο Γιούροβα. Για να δούμε μετά τις ε, ερωτήσεις. colleagues, is everyone ready for the next item for Mrs. Everyone settled and ready. Thank you. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε τώρα στο σημείο 12, το διαρθρωμένο διάλογο με την ε, Επίτροπο Γιώροβα, αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, ε, εσωτερικών και ισότητας των φύλων. Πρόκειται για διαρθρωμένο διάλογο. Καλό λοιπόν είναι να τον διαρθρώσουμε Καλά. Πρώτα θα ακούσουμε τους συντονιστές και μετά τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Θα μιλήσουμε για τις προτεραιότητες για το 2017, το πρόγραμμα εργασιών για το 2016. Και για να μην χρονοτριβούμε θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην Επίτροπο και μετά θα ακούσουμε, επαναλαμβάνω, πρώτα τους συντονιστές και μετά τα μέλη. Δεν είναι πολύ ακόμη στην αίθουσα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα καταφτάσουν κι άλλοι και θα έχουμε μακροσκελή κατάλογο ομιλητών. Οπότε για να έχουμε χρόνο για συζήτηση θα παρακαλούσα την Επίτροπο να είναι συνοπτική στην πρώτη της παρουσίαση για να έχουμε χρόνο για τη συζήτηση και την υποβολή ερωτήσεων. Γιατί είναι πολλά τα ενδιαφέροντα θέματα. Δεν θα περιμένουμε τους συναδέλφους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα και στο μεταξύ θα έρθουν. Κυρία Γιώροβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα καταρχήν να σας ε, συγχαρώ θερμότατα για την επανεκλογή σας στη θέση του Πρόεδρου της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Προσβλέπω σε στενή συνεργασία και φέτος. Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πολλά έχουν μεσολαβήσει και χαίρομαι που σήμερα θα σας ενημερώσω για τις εξελίξεις και θα ακούσω τα σχόλια και τις προτάσεις σας για τη μελλοντική μας συνεργασία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το 2016 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η καλύτερη μας αντίδραση είναι να ε, προετοιμαστούμε καλά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, να ενισχύσουμε την ασφαλειά τους και να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις, ε, τη ρητορική μίσους ε, και το ρατσισμό. Έχουμε πρόοδο σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την καταπολέμηση τη απάτη κατά του δημοσιονομικού του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα δικονομικά δικαιώματα και προχωρούμε σε ό,τι αφορά τη σύσταση τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την στήριξή σα και την επικοδομητική σα κριτική, γιατί χάρη σε αυτά υλοποίησαμε του στόχου μα και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη πυγμή και αποφασιστικότητα και στο δεύτερο ημισή των θητιών μας. Έχουμε μια, ένα στιβαρό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη σωστή του εφαρμογή. Μέσω των κανόνων που υπάρχουν και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Κομισιόν συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις για να υπάρχει σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης ε, καθώς πλησιάζουμε στον Μάιο του 2018. Έχουμε συχνές συναντήσεις με τα κράτη-μέλη και την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για να υπάρξει μια ενιαία εφαρμογή. Ξέρετε ότι πάντα λέω ότι με την υιοθέτηση του γενικού κανονισμού δεν σταμάτησε αλλά ξεκίνησε η υπόθεση αυτή. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας ε, μαζί με τους εταίρους μας ε, και με την Επιτροπή του Άρθρου 29 για να ζωντανεύσει πραγματικά αυτή η υπόθεση και να προχωρήσουμε στον στόχο μας ε, να έχουμε δηλαδή ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ε, πρόταση για την ιδιωτική ζωή αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου Άνσιπ θα ήθελα να πω πως στόχος μας ήταν να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει αντίφαση μεταξύ του γενικού πλαισίου ή αλληλεπικάλυψη μεταξύ του γενικού πλαισίου και των κανόνων ηλεκτρονικής ιδιωτικής ζωής για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού 45 του 2001 έχει στόχο τον εξυγχρονισμό των ε, κανόνων που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα φορείς και αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε στο δυνατόν περισσότερο τα πράγματα με τον γενικό κανονισμό προστασία δεδομένων και οι δύο κανονισμοί θα πρέπει να ισχύουν από τον Μάιο του 2018 μαζί με το γενικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξω εδώ πέρα την ε, στήριξή σας ε, για τις διαπραγματεύσεις επί του κειμένου. Στις 10 ε, Ιανουαρίου η Κομισιόν επίσης παρουσίασε την στρατηγική της προσέγγιση για τις διεθνείς μεταφορές προσωπικών δεδομένων και για την εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών παγκοσμίων. Στόχο έχουμε να διασφαλίσουμε πως όταν μεταφέρονται τέτοια δεδομένα διεθνώς προστασία θα μεταφέρεται μαζί τους. Θέλουμε να συνεργαστούμε με χώρες που θέλουν να έχουν ένα εύρωστο τέτοιο νομικό καθεστώς ε, και κάποιες αρχές προστασίας δεδομένων που θα ανταποκρίνονται στα, ε, σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και βεβαίως θα ξεκινήσουμε ε, συζητήσεις με εμπορικούς εταίρους στην Ασία, ξεκινώντας από την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, οι οποίες πρόσφατα υιοθέτησαν την σχετική τους νομοθεσία. Επιπλέον, θα παίξουμε έναν πιο ενεργό ρόλο στα διεθνή φόρα για να επιτύχουμε υψηλές προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων. Παγκοσμίω, παραδείγματο χάρη, θα ζητήσουμε γρήγορη έγκριση της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στον τομέα της επιβολής του νόμου χρειαζόμαστε ασφαλείς ανταλλαγές προσωπικών δεδομένων που θα βασίζονται σε ισχυρές προδιαγραφές, ε, η συμφωνία Ομπρέλα με τις ίπα που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία τον Δεκέμβριο είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς η συνεργασία των διοκτικών αρχών με ένα σημαντικό διεθνή εταίρο μπορεί να ενισχυθεί με ισχυρές προδιαγραφές. Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως μετά τους διορισμούς ε, των και τους ορισμούς των ΙΠΑ με τη σχετική του νομοθεσία η Συμφωνία Ομπρελά θα τεθεί ενισχύ τον Φεβρουάριο και έτσι οι πολίτες ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν ίση αντιμετώπιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τους στις ΙΠΑ. Σε σχέση με την ασπίδα της ιδιωτικής ζωής θα ήθελα να σε ενημερώσω πως η Κομισιόν και οι αρχές μας ε, προστασίας των προσωπικών δεδομένων συνεργάζονται στενά με τις ΙΠΑ. Αυτή τη στιγμή 1.700 εταιρείες έχουν έγγραφη και το σύστημα λειτουργεί επαρκώς και τώρα βασίζομαι στην νέα Αμερικανική κυβέρνηση για να διατηρήσει τις δεσμεύσεις που αποτελούν την βάση αυτής της ασπίδας της ιδιωτικής ζωής. Αυτό σημαίνει να διατηρηθεί η Προεδρική Οδηγία Υπαριθμών 88 που είναι ε, η βάση της ασπίδας για την ιδιωτική ζωή και αφορά την επιπρόσθετη πρόσβαση για λόγους εθνικής ασφαλείας στα στοιχεία αυτά, καθώς επίσης και να λειτουργεί επαρκώς η νέα υπηρεσία συνεγόρου του πολίτη. Επίσης, οι αρμόδιες ε, ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές θα εμπλακούν στην κατάρτιση της νέας συμφωνίας και έχω ήδη πει πώς ενδιαφέρομαι για να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Αλλά, ακόμα και μετά την πρώτη κοινή αναθεώρηση, θα έρθω σε επαφή με τους Αμερικανούς ομολόγους μου για να τονίσουμε την ανάγκη πλήρους εφαρμογής από την πλευρά των ΗΠΑ και σκοπεύω να επισκεφτώ τις ε, ΗΠΑ στην, την Άνοιξη. Τώρα, να αναφερθώ λίγο στα ζητήματα ποινικού δικαίου. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για την στήριξή σας, για την ε, οδηγία καταπολέμησης της απάτης. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ε, κοινότητας για την καταπολέμηση της σοβαρής διασυνοριακής απάτης ε, ΦΠΑ που θα περιληφθεί έτσι στην οδηγία και άρα σε αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής εισαγγελία. Ε, πλέον αλλάζουν τα πράγματα, ουσιαστικά θα έχουμε έτσι μια ουσιαστική αντίδραση για να καταπολεμήσουμε τέτοια πολυπλοκά εγκλήματα. Πριν από ένα χρόνο κανείς δεν πίστευε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και τώρα έχουμε τις μεγάλες διασυνοριακές τι ΦΠΑ που έχουν μπει στην οδηγία αυτή. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στόχος μου είναι και ήταν πάντα να υπάρξει μια ανεξάρτητη και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά το οποίο θα έχει τα μεγαλύτερα ωφέλη για τον κοινό μας προϋπολογισμό και για τον χώρο ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύνης. Όμως το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης του Δεκεμβρίου η Σουηδία δήλωσε ότι δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η έλλειψη ομοφωνίας ε, επιβεβαιώθηκε και από το Κορεπέρ την προηγούμενη εβδομάδα. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης θα συναντηθούν την Παρασκευή σε άτυπο Συμβούλιο για να συζητήσουν το ζήτημα και τα επόμενα βήματα. Εάν το Συμβούλιο πράγματι δεν καταφέρει να φτάσει σε ομοφωνία, η συνθήκη προβλέπει πως οι χώρες που είναι διατεθειμένες να ξεκινήσουν την υπηρεσία μπορεί να παραπέψουν το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βασίζομαι στην πλήρη στήριξή σας ε, για την σύσταση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ακόμα και υπ' αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Οι μου συνεργάζονται με την Προεδρία της Μάλτας, έτσι ώστε να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να είμαι ξεκάθαρη, η Εισαγγελία απαιτεί την συμμετοχή σημαντικού αριθμού κρατών μελών. Τον Δεκέμβριο η Κομισιόν πρότεινε έναν κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των ε, διαταγών αναγκαστικής ε, εκτέλεσης και κατάσχεσης ε, και έτσι δεν θα μπορούν οι εγκληματίες να κρύβουν τα περισσότερα στοιχεία σε άλλα κράτη-μέλη. Πάνω από το 98% των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κατασχεθούν αν υπάρχει διασυνοριακό ζήτημα. Η πρόταση θα αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα και προτείνουμε κανόνες που θα εφαρμόζονται άμεσα με σύντομε προθεσμίες για διαταγές παγώματος των παρισιακών στοιχείων. 48 ώρες για αναγνώριση και εκτέλεση εντάλματος με βάση τυποποιημένα έντυπα. Ένα άλλο περίπλοκο ζήτημα που μα απασχολεί είναι η διασυνοριακή πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα, έχει όμως σύνορα η δικαιοδοσία των κρατών μελών. Οπότε, όπως ζήτησε και το Συμβούλιο, εργαζόμαστε σε μία συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Υπάρχει βεβαίως και το θέμα της πρόληψης ε, της χρηματοδότησης τρομοκρατικών και εγκληματικών δραστηριοτήτων και έχουμε και την προτινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος. Όπως ξέρετε ε, υπάρχει μια εντολή του Συμβουλίου και ελπίζω να ακολουθήσει σύντομα και το Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα ή αν όχι αυτή την εβδομάδα το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά την διαφάνεια του τελικού δικαιούχου. Να πω επίσης πώς άκουσα τις ανησυχίες σας ε, που εκφράσατε την προηγούμενη εβδομάδα στην ε, πράξη κατεξιοδότηση για τις ε, τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Το παίρνω πολύ στα σοβαρά και ετοιμάζουμε μία αξιολόγηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν την καταπολέμηση των δικαιωτικών μεταχειρήσεων και των λόγων μίσους, καθώς επίσης και τη μεταχείριση των Ρωμά. Λοιπόν, να δούμε τον κώδικα συμπεριφοράς ε, που συμφωνήσαμε με κάποιες εταιρείες τον Μάιο του 2016. Είχαμε κάποια πρόοδο, αλλά βεβαίως υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Βεβαίως ε, υπήρχαν διαφορές ανάλογα με το κράτος ε, μέλος και με το κατέβασμα παρανόμων σελίδων. Τα αποτελέσματα βέβαια εξαρτώνται και από την σελίδα ή την χώρα όπου είχαμε τις ε, κινητοποιήσεις, κάτι το οποίο βεβαίω δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Κοιτάμε επίσης και πρόοδο σε άλλους τομείς όπως η διαφάνεια απέναντι στους χρήστες και το θέμα θετικών αφηγημάτων με θετικά αφηγήματα ή αντιαφηγήματα από την κοινωνία των πολιτών μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο κατά της ριζοσπαστικοποίησης και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καθώς αναφερθήκατε στο φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού και συγκεκριμένα για την προστασία των παιδιών ε, στην μετανάστευση. Έχουμε την χρηματοδότηση της Δάφνης ε, που το 2016 αφορούσε αυτό το ζήτημα και ετοιμάζουμε μια κοινή ανακοίνωση για το σχέδιο δράσης για τους ασυνόδευτούς ανηλίκους. Ε, ανακοινώνουμε νέες δράσεις ε, και συστάσεις προς τα κράτη-μέλη και μας αποσχολεί και το ζήτημα των γυναικών μεταναστών, το πώς ε, επίσης ε, θα αναγνωρίζουμε τα ευπαθή άτομα που ετούνται άσυλο και παρέχουμε χρηματοδότηση για να στηριχθεί η ένταξη των γυναικών προσφύγων. Όπως ξέρετε, προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κυρώσει την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία περιέχει διατάξεις που αφορούν τις ε, μεταναστρίες. Και αναμένουμε περαιτέρω δράση στον τομέα αυτών. Δεν θα πρέπει να συνεχιστούν οι διακρίσεις. Ιδιαίτερα στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό και στηρίζουμε τα κράτη-μέλη, ενώ ταυτόχρονα ε, ξεκινήσαμε και διαδικασίες επί παραβάση στα πλαίσια της οδηγίας της φιλητικής ισότητας και στα πλαίσια της οδηγίας πλαίσια του Συμβουλίου για το, για το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Και μάλιστα φέτος ε, θα ξεκινήσουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου των εθνικών στρατηγικών Κοινωνική ένταξης των Ρωμά. Έτσι θα ξεκινήσει η διαδικασία για να προετοιμάσουμε τη στρατηγική μετά το 2020, τότε που θα λήξει το ισχύον πλαίσιο στρατηγικής. Επίσης εφαρμόζουμε ένα κατάλογο δράσεων υπέρ της ισότητας των ΛΟΑΔΜ. Σας υποβάλαμε το σχετικό κατάλογο δράσεων πέρυσι και μάλιστα το Φεβρουάριο θα λάβουμε μέρο σε μια διάσκεψη τη Μαλτέζική Προεδρία και θα σα ενημερώσουμε περαιτέρω για την εφαρμογή αυτού του καταλόγου δράσεων. Επίση, θα ήθελα ολοκληρώνοντα να υπογραμμίσω την ανάγκη, τη σημασία που έχει η στενή μα συνεργασία σε όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και μάλιστα να τα ενισχύσουμε προκειμένου να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Περιμένω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας για το πώς θα υλοποιήσουμε αυτούς τους κοινούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μας υπενθυμίσατε την πληθώρα των ζητημάτων που είναι όλα πολύ σημαντικά και, και σήμερα αλλά και αύριο στο διαρθρωμένο διάλογο με τον Επιτροπό Αβραμόπουλο ε, θα επισημάνουμε πολλά θέματα και σήμερα και αύριο, αύριο λιγότερα, αλλά είναι όλα ε, εξίσου σημαντικά και φλέγοντα και ίσως θα πρέπει ε, να έχουμε και άλλες συναντήσεις για να επισέλθουμε πιο αναλυτικά στα επιμέρους θέματα, γιατί δεν μπορούμε μέσα σε μια μέρα να καλύπτουμε τόσο μεγάλη γάμα θεμάτων. Ίσως θα πρέπει, θα πρέπει να δούμε έναν τρόπο για το πώς πιο διεξοδικά μπορούμε να, και εμπεριστατωμένα να επιληφθούμε αυτό το θεμάτων. Εν πάση περιπτώσει, επικεντρωθούμε στα βασικά ζητήματα. Θα ξεκινήσω, όπως είπα, με τους συντονιστές μας και τους θερμοπαρακαλώ να μην υπερβούν το δίλεπτο γιατί είναι εκτενέστατος ο κατάλογος και για να προλάβουν να μιλήσουν όλοι πρέπει να περιοριστούμε στο χρόνο μας. Θα ακούσουμε τους συντονιστές, θα υποβάλλουν τι ερωτήσεις, θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο για τις απαντήσεις και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπους βουλευτές. Ξεκινούμε από, το, από τη συντονίστρια του ΕΛΚ, την κυρία Μετσόλα. Ευχαριστώ, Κλώτ, και ευχαριστώ την Επίτροπο. Θα είμαι λακωνική για να μπορέσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να θέσουν τι ερωτήσεις του. Αναφέρατε το, τη δύσκολη χρονιά που είχαμε πέρυσι, το 2016 Θέλω κάποιες επιβεβαιώσεις όμως, κάποιες διαβεβαιώσεις για το κατά πόσο είχατε απόλυτες δεσμεύσεις και, δείξεις από, και δείξει από τις από τα κράτη-μέλη μάλλον θα τηλήσουν τις υποχρεώσεις τους και τις Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο. Είπατε για την, αυτή τη Γενική Συμφωνία, την ασπίδα της ιδιωτικής σφαίρας, της ιδιωτικής ζωής. Ε, τι δεσμεύσει έχουμε από τι ΗΠΑ ώστε οι συμφωνίε αυτέ να εφαρμοστούν και εμπράκτο. Επίση, αναφερθήκατε στι συμφωνίε προστασία δεδομένων με άλλε χώρε όπω την Ιαπωνία. Τι γίνεται με τι άλλε υπήρου, πώ ε, προχωράνε οι συζητήσει εκεί, άσχετα με τι εθνικέ του ε, νομοθεσίε για την προστασία των δεδομένων. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ε, των ευάλωτων μεταναστεριών τι δράσεις ε, θα αναλάβετε πέραν της απλής χρηματοδότησης και το κονδύλιο που θα δώσετε στα κράτη-μέλη που χρειάζονται ε, τέτοια μέτρα για τη στήριξη των γυναικών ευάλωτων. Η κυρία ε, Ζίπελ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Γιώροβα. Θα υποβάλω κάποιες ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. έχω μεγάλε αμφιβολίε αν θα στεφθεί με επιτυχία μια τέτοια πρωτοβουλία αν δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Και ακόμη κι αν συμμετέχουν, ποια θα είναι τα συγκεκριμένα δικαιώματα και οι εξουσίες αυτής τη Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε σχέση με τις εθνικές εισαγγελικέ αρχές και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλή συνεργασία μεταξύ του, Γιατί αν δεν έχουμε σαφείς εξουσίε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, ποια θα είναι ε, τα αποτελέσματα, οι συνέπειες στους υπόπτους ή τους κατηγορουμένους και στα δικά τους δικονομικά δικαιώματα. Δεν θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να αναπτύξουμε περαιτέρω το ποινικό δικονομικό δίκαιο και πέραν του πρώτου πακέτου για, τα, για τις δικονομικές διατάξεις. Δεύτερον, τι γίνεται σε ό,τι αφορά το παραδεκτό των αποδείξεων, των τεκμηρίων, γιατί και εκεί είναι διαφορετική κατάσταση στα κράτη-μέλη. Δεν χρειαζόμαστε και για τις αποδείξεις αφής κανόνες. Έχω και μια άλλη ερώτηση. Ε, έχουμε ε, βάσει δεδομένων ε, και μιλούμε πολύ συχνά για προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτές όμως οι βάσεις δεδομένων όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου. Οπότε τι δικονομικές εγγύησεις έχουμε, όπως το τεκμήριο της αθωότητας, ε, ισχύουν όλα αυτά, όλες αυτές οι δικονομικές εγγύησεις στις διαδικασίες χρήσης των δεδομένων. Επίσης, τι γίνεται στις συζητήσεις για την διαλειτουργικότητα. Και τέλος, συνεχίζονται οι συζητήσεις, όχι μόνο σε μία-δύο χώρες, ε, συζητήσεις που δείχνουν ότι επιδεινώνεται η κατάσταση των γυναικών και καταπατώνται τα δικαιώματά τους. Προτείνεται να αναλάβετε περαιτέρω το πρωτοβουλίο σε αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, ε, το Συμβούλιο της Παρασκευής ε, θα μιλήσει για αυτά τα θέματα. Κυρία Ιντβελτ, ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε κυρία Επίτροπε. Εν συντομία, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Τι γίνεται με τη διατλαντική κατάσταση. Η συμφωνία ομπρέλα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, δεν κάνω λάθος. Προϋπόθεση όμως για την ε, εφαρμογή της είναι οι εξαιρέσεις από το νομοσχέδιο για την ιδιωτική σφαίρα να ε, αποσυρθούν. Τι έχει εγγυηθεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου και αν δεν γίνει, ε, ποια θα είναι η κατάσταση. Κατά την γνώμη μου δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί, δεν θα είναι έγκυρη η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά την ασπίδα για την ιδιωτική ζωή. Η διαμεσολαβήτρια έχει αποχωρήσει, αλλά δεν έχει διοριστεί ακόμη νέος διαμεσολαβήτης. Τι και έχουμε ότι ο νέος διαμεσολαβητής, παρόλο που δεν έχω πιστεί για την ε, ιδιότητα αυτή, ότι θα ε, οδιοριστεί εγκαίρος. Και μάλιστα ο πρώην πρόεδρος ε, Ομπάμα πριν να αποχωρήσει είχε, επιτρέψει, είχε υιοθετήσει κάποιους κανόνες για την διαχείριση των δεδομένων από την NSA. Ε, θεωρείτε ότι αυτοί, αυτοί οι κανόνες συνάδουν με τη συμφωνία για την ασπίδα για, για την ιδιωτική σφαίρα. Επίσης, ε, με προβληματίζει η στρατηγική προσέγγιση για τη μεταφορά δεδομένων, μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται ως βασική μας εμπορική εταίρη. Και αν ε, οι διαπραγματεύσεις που, έχουμε, που είχαμε με τις ΗΠΑ για τη διατλαντική μεταβίβαση δεδομένων δεν ευωδόθηκε, ε, φοβάμαι ότι δεν θα υιοθετηθούν οι ίδιε προδιαγραφές σε όλε αυτέ τι συμφωνίε και πάλι για τη συμφωνία αυτή τη γενική, την συμφωνία Ομπρέλα και τις εξαιρέσεις από την Privacy Act, από το νομοσχέδιο, από το νόμο των ΗΠΑ για την ιδιωτική σφαίρα. Και τι γίνεται με τις συμφωνίες για το PNR και το SWIFT και την ετήσια αναθεώρηση. Χαίρομαι επιτέλους που υποβλήθηκαν αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης, γιατί τις περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Επίσης, αυτές οι δύο συμφωνίες εξαιρούνται από την συμφωνία για την ιδιωτική σφαίρα και τι αντίκτυπο έχει κάτι τέτοιο στη δική του εγκυρότητα. Γιατί λέμε ότι η συμφωνία ομπρέλα, γενική αυτή η συμφωνία, θα είναι έγκυρη αν καταργηθούν αυτέ οι εξαιρεσει. Οπότε λείπουν ακόμη σημαντικά ε, στοιχεία. Και δεν ε, είμαι σίγουρη ότι ο πρώτος ΤΑΜ θα είναι ο νέος ε, πρωτεργάτης ε, της προστασίας των δεδομένων, ο νέος πρωταθλητής στην προστασία των δεδομένων, εκτό και αν έχετε κάποια στοιχεία περισσότερα εσεί. Ουδέν σχόλιο για το τελευταίο ζήτημα. Κυρία Σαργεντίνη, σας ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις έχω να υποβάλω. Ερώτηση πρώτη. Φαίνεται ότι πέρασε πολύ καιρό, αλλά την περασμένη εβδομάδα τελευταία μέρα της Προεδρίας του, ε, ο πρόεδρος Ομπάμα επέτρεψε στην NSA να δώσει τα στοιχεία που είχε και σε άλλες υπηρεσίες όπως τη CIA, την FBI και το καθεξής. Αυτές είναι πληροφορίες από την New York Times ποιες θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης ε, στην ασπίδα για την ιδιωτική σφαίρα. Γιατί μέχρι στιγμής η NSA ε, μπορούσε να μοιράσει την, ανάλυση της άλλης μυστικής υπηρεσίας, αλλά όχι τα στοιχεία καθε αυτά. Οπότε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα της ισότητας και της πάταξης των διακρίσεων. Πέρυσι ε, είχε κυκλοφορήσει αυτό το εγχειρίδιο για την ισότητα και με τους ΛΟΑΔΜΟ και εγώ και η συνάδελφος ε, Ολύρη και Λούνα Τσέκ να μαθ θέλουμε να μάθουμε τι συνέχεια δόθηκε σε αυτόν τον οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των ΛΑΔΜΑ. Γιατί μας υποσχεθήκατε τακτικές εκθέσεις πρόοδου για τα θέματα των ΛΟΑΔΜ. Τι έγινε πέρυσι από την υιοθέτηση του καταλόγου δράσεων και σε ό,τι αφορά την ε, οδηγία για την ε, ίση μεταχείριση την επιστολή ανάθεση καθηκόντων ο πρόεδρος Γιουνκέρα σας ε, ε, ανέθεσε την, ε, το θέμα αυτό και μάλιστα ανέλαβε δέσμευση, να υλοποιήσει τη δέσμευση του 2009. Εν ώψη και της Μαλτέζικης Προεδρίας σκοπεύεται να λάβετε συγκεκριμένες δράσεις του τους, επόμενους, τους επόμενους μήνες για να ξεμπλοκάρετε επιτέλους αυτή την οδηγία για την ίση μεταχείριση. Ευχαριστώ. Επίτροπε, να απαντήσετε και θα ήθελα να μου δώσετε ε, το κείμενο του ε, Γενικού Εισαγγελέα ε, για τις δικαιούχες χώρες. Δεν θα δώσω το λόγο στους συντονιστές που δεν είναι εδώ. Υπάρχουν τόσοι πολλοί βουλευτέ που θέλουν το λόγο. Γι' αυτό θέλω να προχωρήσουμε, ούτω ώστε όλοι όσοι είναι παρόντες να έχουν χρόνο να μιλήσουν. Απαντήστε λακωνικά, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ομιλητέ που περιμένουν, πολλούς ε, βουλευτές που περιμένουν να μιλήσουν. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις ε, ε, τι γίνεται ε, με τα θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ μετά την αλλαγή της κυβέρνησης, του Πρόεδρου. Ε, καταρχάς, για θέματα ιδιωτική σφαίρα και της ασπίδας. Ξέρετε πολύ καλά ότι η λειτουργία της ασπίδας αυτής είναι μία ε, διαδικασία, δεν είναι μία απόφαση που την παίρνουμε και τελείωσε. Το σύστημα είναι ένα μηχανισμό ο οποίος προβλέπει πολύ αξιόπιστες ε, και συνεχείς δράσεις και την υλοποίηση διαφόρων υποχρεώσεων και από τις δύο πλευρές. Η βασική υποχρέωση είναι εμπίπτει βέβαια στο γήπεδο των Αμερικανών. Έχουμε 7 φορείς, κρατικούς φορείς, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξεκίνησαν με βάση τη συμφωνία για την, προστασία, για την ασπίδα της ιδιωτικής σφαίρας. Έχουμε την Ομοσπονδιακή Επιτροπή για το Εμπόριο. Έχουμε τους φορείς ε, κρατικής ασφάλειας, οι οποίοι θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Εγώ περιμένω συνέχεια μετά την ανάληψη των καθηκών του νέου Προέδρου. Δεν μπορώ να προβλέψω από τώρα ή να πω ότι ο κύριος Τραμπ, ας πούμε, θα είναι ο πρωταθλητής ή δεν θα είναι ο πρωταθλητής, ας πούμε, ε, της ιδιωτικότητας ε, των Ευρωπαίων. Κανένας μας δεν μπορεί να το πει αυτό. Όμως, εγώ ήρθα σε επαφή με τους ε, ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στην Αμερική, με την ομόλογό μου στις διαπραγματεύσεις με, μίλησα με βουλευτές, με έναν ευρωβουλευτή που έστειλε μια επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ ε, και του εξήγησε τη σημασία της διασφάλισης αυτής της ασπίδας. Και, τη και την προστασία των δεδομένων ε, των Ευρωπαίων που πηγαίνουν από την Ευρώπη στην Αμερική. Σκοπεύω βεβαίω να μεταβώ στι ΗΠΑ και εγώ το συντομότερο δυνατόν, τον Απρίλιο κατά πάσα πιθανότητα, να συναντήσω του ομολόγου μου, που, τον ομολόγο μου που θα είναι ο κύριο Ρο, για να συζητήσω και με εκείνον, αλλά και με, την, ε, με μια αντιπροσωπεία ε, για θέματα ασφάλειας και να τονίσω την απόλυτη σημασία, απόλυτη προτεραιότητα ε, που έχει για μας αυτή η ασπίδα και ότι πρέπει να διατηρηθεί συνέχεια. Αλλιώς θα πω ότι πρόκειται για μονομονεμερή απόφαση η οποία ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μπορεί να ανασταλεί με μονομερή απόφαση. Αυτό σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το σύστημα. Παρακολουθούμε τι γίνεται με την προοδική οδηγία 28 που είναι βασικός πυλώνας στην Αμερικανική νομοθεσία και παρακολουθούμε και τι θα κάνει η Αμερικανική πλευρά με άλλα νομοθετήματα, το πώς θα υλοποιήσει όλες τις προϋποθέσεις που απαγορεύουν τις μαζικές παρακολουθήσεις και που αφήνει τη δυνατότητα συλλογής δεδομένων μόνο υπό τις προϋποθέσεις της ανάγκης και της αναλογικότητας. Μόνο εφόσον υπάρχει ανάγκη λοιπόν και υπάρχει αναλογικότητα. Παρακολουθούμε λοιπόν τα τεκτενόμενα στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Και φυσικά θα ρωτήσουμε πολύ σύντομα τους Αμερικανούς τι θα γίνει με τη θέση του διαμεσολαβητή. Δημιουργήθηκε αυτή η θέση ε, για να εξυπηρετήσει την ασπίδα για την ε, ιδιωτικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ασχοληθεί με κανένα παράπονο ακόμη παραβίαση της ιδιωτικότητας. Επίσης, εγώ θα ήθελα κάποιος ε, επιπλέον να ξεκινήσει, ας πούμε, να κάνει τον αρθήρο λάκτισμα και να κάνει ένα παράπονο και να το απευθύνει προς τον διαμεσολαβητή μέσω του Twitter. Θα δούμε ε, υπάρχει ανεξαρτησία από το, τους φορείς ε, εθνικής ασφάλειας και ανεξαρτησία γενικά ε, της θέσης αυτής του Διαμεσολαβητή. Και ανεξαρτησία από τον Υπουργό βεβαίω. Εξωτερικών. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τον Τραμπ και που λένε ότι είναι επιχειρηματίας, που καταλαβαίνει πολύ καλά το πώς λειτουργεί το εμπόριο και επιχειρήσεις, ας πούμε, ε, και τι εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις. Εγώ θα πω στους Αμερικανούς εταίρους ότι εμείς θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, το τι κάνουν οι Αμερικανοί, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων. Θα συλλέγουμε τα δεδομένα για την πρώτη ετήσια έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί ε, το Σεπτέμβριο. Έχουμε διάφορα κανάλια, όχι μόνο τις πληροφορίες από τις επίσημες αμερικανικές πηγές, αλλά και από, το, από διάφορες εποπτικές αρχές, watchdog, από τον τύπο και δημοσιεύματα του τύπου. Και φυσικά έχουμε και τις δικές μας προστασί... ε, υπηρεσίες προστασίας δεδομένων που παρακολουθούν και αυτές την κατάσταση. Η πρώτη ετήσια επισκόπηση θα έχει λοιπόν θα είναι η απεικόνηση της πραγματικότητας με στοιχεία. Δεν θα υπάρχει καμία, εξο, ένα, κανένας εξοραϊσμός της κατάστασης. Και οι Αμερικανοί θα καταλάβουν πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει την προστασία των δεδομένων των Ευρωπαίων για την ε, συμφωνία πλατφόρμα, «Πλατφόρμα-Ομπρέλα». Στις 17 Ιανουαρίου του 2017, ο Γενικός εισαγγελέα. Ε, διόρισε διάφορα άτομα, παραδείγματο χάρη στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, και στο FBI, ας πούμε, άτομα και στην κοινοποίηση προς το Συμβούλιο, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, εξήγησαν ότι με αυτούς τους διορισμούς έχουν ολοκληρώσει τις εσωτερικές διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας και επομένως η συμφωνία τίθεται σε ισχύ 1η Φεβρουαρίου, όπως είπα και προηγουμένως. Εάν χρειαστεί στο μέλλον να υπάρξουν και πλέον ε, υπηρεσίες, δηλαδή αν η νέα κυβέρνηση αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο στο, στην Αμερικανική νομοθεσία, τότε έχουμε δεσμευτεί η κοινοποίηση αυτή να αναφέρει και αυτές τις μάλλον κοινοποίηση να αναφέρει και αυτές τις νέες υπηρεσίες. Είναι μια διαδικασία, δηλαδή, εν εξελίξη. Δεν είναι μια απόφαση που παίρνετε εν μια νυχτή, ας πούμε, και τελειώνει εκεί. Αυτή είναι η κατάσταση. Η δήλωση θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα 1η Φεβρουαρίου, μαζί με την επίσημη αναγγελία για τη θέση ισχύ λοιπόν της συμφωνίας. Η δήλωση έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου όταν υιοθετήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου για να ολοκληρωθεί η Συμφωνία Ομπρέλα στις 2 στις 2 Δεκεμβρίου του 2016. Οι διεθνείς μεταβιβάσεις, μεταφορές, ε, διότι της κυρίας Ιντβέλτ. Αναγγείλαμε ότι θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αποφασίσουμε στο μέλλον με άλλες αποφάσεις ε, του Συμβουλίου σε περίπτωση που κάποια τρίτη χώρα έχει τις απαραίτητες διασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των ανθρώπων Μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου στην υπόθεση ΣΡΕΜΣ μίλησε για ξεκάθαρα κριτήρια για να βασίζεται αυτή η απόφαση επάρκειας ε, και αναφέρει και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται. Αυτή είναι η βασική μας αρχή. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή με την Ιαπωνία και με την Νότια Κορέα, όπου έχει υιοθετηθεί εκεί η νομοθεσία πρόσφατα για να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων και μεταξύ των τρίτων χωρών υπάρχουν 108 χώρες που έχουν μια κάποια νομοθεσία που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, αλλά μόνο κάποια από αυτά τα κράτη είναι οι πιθανοί υποψήφοι, ούτως ώστε να για παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασής τους ούτως ώστε να αρχίσουμε να σχεδιάσουμε την απόφαση επάρκειας. Ξέρετε ότι μια τέτοια απόφαση επάρκειας ενέχει και κινδύνους. Κινδύνους που πρέπει να δεχτεί η Κομισιόν. Γιατί σε κάποιο βαθμό γινόμαστε συνυπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στην τρίτη αυτή χώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επίσης, θέλουμε να παρακολουθούμε στη Βραζιλία πιο πολύ την κατάσταση και για την Ασία έχουμε στο μυαλό μας την Ινδία στο μέλλον. Αλλά για φέτος θα εργαστούμε πολύ πιο έντονα για να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στην τρίτη χώρα και αυτές οι ξένες χώρες είναι η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Για τις, εσωτερι... για τις βάσεις δεδομένων και για τη γαλλιτουργικότητα των βάσεων δεδομένων έχετε απόλυτο δίκιο ότι είμαστε πολύ δραστήριοι. Μας, αναγκάζει... Μας αναγκάζουν και οι απειλές στην ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε και η ανάγκη να γνωρίσουμε καλύτερα το ποιο, άτομα κινούνται στις ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ε, εφαρμόζουμε το σύστημα SIS, ε, ετοιμάζουμε το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου, ετοιμάζουμε και άλλα συστήματα τα οποία λειτουργούν με συλλογή προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων, υπηκών τριτών χωρών, Και εμεί από πλευρά Κομισιόν ψάχνουμε να βρούμε πάντα τον καλύτερο τρόπο για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των ανθρώπων και εμπλεκόμαστε στη δουλειά που κάνουν, που γίνονται για αυτά τα νέα ή παλιά συστήματα. Και ούτως ή άλλως αν δεν επικυρώσουμε εμείς αυτά τα συστήματα, αν δεν δώσουμε το πράσινο φως, κανένα από αυτά δεν μπορεί να, ούτε να προταθεί ούτε να αρχίσει να λειτουργεί. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία 100% και συνδιαμορφώνουμε τα υψηλά ε, πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Το δεύτερο που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι η διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών και η καλή λειτουργία τους. Γιατί όλα αυτά είναι εκδοτικά συστήματα φυσικά είναι και πολύ δαπανηρά μεταξύ άλλων και θα πρέπει να λειτουργούν με τον καλύτερο ε, και πιο οικονομικό τρόπο. Για το γραφείο της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, χάσαμε την ομοφωνία με την αναγγελία της Σουηδίας Επίσης, ε, είδαμε τι έγινε στην ψηφοφορία στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο, το οποίο απέρριψε την πρόταση, ή τουλάχιστον δεν συμφώνησε η Ολλανδία να γίνει η έδρα του μελλοντικού, της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Η Πολωνία και η Ουγγαρία είναι υποψήφοι. Πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα, λοιπόν. Εγώ έχω ε, επισκεφθεί αυτές τις χώρες και τα εθνικά τους κοινοβούλια. Είμαι σε επαφές με τους υπουργούς δικαιοσύνης των χωρών αυτών. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι χώρες αυτές θέλουν να μείνουν στο περιθώριο του συστήματος αυτούς, για διαφορετικούς λόγους. Να σας πω ποια είναι η λογική και η επιχειρηματολογία των Σουηδών. Άκουσα από διάφορους ε, βουλευτές Σουηδούς ότι η Σουηδία δεν χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί η δική του εισαγγελία λειτουργεί θαυμάσια. Κάποια παρεξήγηση υπάρχει εδώ, έτσι. Γιατί εμεί δεν δημιουργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να βελτιώσουμε την εισαγγελία στα κράτη-μέλη, έτσι. Δημιουργούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να ενισχύσουμε τι εθνικέ εισαγγελίε. Για να καταπολεμούν καλύτερα τα εγκλήματα ε, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν αυτές οι χώρες μείνουν στο περιθώριο, παρετούνται ουσιαστικά από την ευκαιρία να ελέγχονται, να ελέγχεται ο τρόπο με τον οποίο ξοδεύονται τα λεφτά των φορολογουμένων τους. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι η Σουηδία, ας πούμε, ε, συνεισφέρει, είναι καθαρός φορέας των ε, στον κοινοτικό προπολογισμό. Επίσης πήγα στην Πολωνία, μίλησα με τους υπουργού. μίλησα με σημαντικούς ανθρώπους που επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει εκεί ένα συνταγματικό πρόβλημα. Έτσι μου λένε. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα. Αλλά πώς ένα κράτος μέλος το οποίο ε, λαμβάνει το 1 τέταρτο των κονδυλίων των διαφορετικών ταμείων να βγει εκτός από αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα δημιουργηθεί ακριβώς για να ερευνά και να διώκει εγκλήματα απάτης και διαφθοράς ε, κατά των κονδυλίων των διαφορετικών ταμείων. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς γίνεται. Και αν ναι, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πώς θα ε, διαμορφωθεί η νέα πολιτική συνοχή, αν υπάρξει νέα πολιτική συνοχή μετά το 2020. Και θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να είναι ένας ε, συνομιλητής. Επίσης, ό,τι αφορά τη μεγάλη απάτες κατά του ΦΠΑ, τις απάτες τύπου καρουσέλ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Μου δίνει τη δύναμη να πιέσω για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτω ώστε να πιστούν όσο να τον περισσότερα κράτη-μέλη ε, να συμμετέχουν στην ίδρυση αυτού του νέου θεσμού. Η στιγμή αληθείας θα είναι μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το αν θα γίνει ή όχι. Γιατί θα υποβάλλουμε μάλλον το Μάρτιο την απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εκεί θα δούμε πόσα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να προχωρήσουν. Για τις αρμοδιότητες για θέματα γυναικών και μεταναστών. Όχι, θα ήθελα να τα απαντήσετε μετά αυτά τα ερωτήματα. Θα μιλήσω πάλι για τις αρμοδιότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για γυναίκες και μετανάστες. Ναι, η κυρία Ιντβέλτε. Είχα κάνει ένα βασικό θέμα για την ανάκληση των εξαιρέσεων ε, στην, στο Privacy Act. Σας άκουσα προσεκτικά και όμως δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Κοιτάξτε, περιμένουν και άλλοι υπομονετικά να μιλήσουν. Καταγράψτε το παρακαλώ, Επίτροπε, και να απαντήσετε στο τέλος. Θέλω να προχωρήσουμε με τις ερωτήσεις των υπολείπων ευρωβουλευτών. Ένα με δύο λεφτά. Το πολύ, γιατί έχω τεράστιο κατάλογο. Θα σα δώσω το λόγο με, τον με, το... με βάση το ποιο ζήτησε πρώτος το λόγο. Θα είμαι πολύ αυστηρό. Ευχαριστώ, Κλοντ, και συγχαρητήρια και πάλι για το ότι επανεκλεγήκατε, Πρόεδρος, και χαίρομαι που παρά το Brexit ε, υποστηρίζουμε ακόμα τους ε, Βρετανούς, ε, πήγαν από συντηρητικούς εργατικούς ευρωβουλευτές. Λοιπόν, συγχαρητήρια και πάλι. Κύριε Επιτροπέ, έχω μια ερώτηση για σας. Αυτή τη στιγμή οι ευρωβουλευτέ πάνω από 400 από εμά ε, προετοιμάζουμε μια έκκληση για σας για το θέμα του Amber Alert. Αυτή τη στιγμή η τσεχική αστυνομία αναζητά την Μιχάλκα, ένα κοριτσάκι που χάθηκε στο, στην Μπλάνταμ κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, στην Τσεχία. Απαιτείται δράση λοιπόν. Θα μπορούσαμε έτσι να σώσουμε ζωές παιδιών σε πολλές χώρες. Η Μάλτα ήταν μία από τις χώρες που έχει εφαρμόσει αυτό το σύστημα προειδοποίησης. Η Σλοβενία και η Κροατία είναι στην διαδικασία εφαρμογής. Εμείς θα θέλαμε το σύστημα αυτό να λειτουργεί σε ολόκληρη την Ένωση. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να περιληφθεί αυτή η έκκληση στα έγγραφα εργασία σας. Δεν θέλω να προωθήσω κάποια οργάνωση και δεν υποχρεωτικό να συνεργαστείτε με κάποια. Αλλά θα ήθελα να δείτε το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ως κράτη-μέλη στην περίπτωση που χάνονται παιδιά. Νομίζω ένα παράδειγμα από τα πολλά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ε, και δεν θα κάνω άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσενίτση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε εδώ. Θέλω να αναφερθώ στο ε, πακέτο προτάσεων που παρουσιάστηκε στις 21 ε, Δεκεμβρίου για να σταματήσει η χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματο και της τρομοκρατίας. Κυρίως ε, μιλάω για την πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της, αναγνώριση, τη εντολή αναγνώρισης της ε, εντολής παγώματος και δέσμευσης ε, περιουσιακών στοιχείων. Καλό είναι αυτό, φυσικά. Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο νομικό εργαλείο για την αναγνώριση των αποφάσεων ε, δέσμευση και παγώματο περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά η Κομισιόν θα μπορούσε να δείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία. Μετά την εμπειρία τη Ιταλία, η οποία αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα οργανωμένου εγκλήματο και πριν από λίγα χρόνια πολιτική τρομοκρατία ε, και να βασιστώ σε αυτό το μοντέλο. Ακριβώ γι' αυτό σα ρωτάω. Δεν θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλάβετε στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία πάντα σε σχέση με τις ε, εγγυήσεις ε, τις δικονομικές και, τις, ε, και την το προληπτικό πάγωμα, την προληπτική δίμευση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Ειδικά όταν μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα ή μαφιόζικο έγκλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα, γιατί τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μέσω του, της χρηματοδότησης. Επίσης, για τους μη Συνοδευμένου, για τους ασυνόδευτους δηλαδή, ανηλίκους. Θαυμάσια συνεργασία είχαμε με την Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ. Ε, στην ομάδα αυτή είμαστε συμπρόεδροι. Τι άμεσα μέτρα θα θέσει η Κομισιόν για να προστατεύσει τους ασυνόδευτους ανήλικους ε, που το νούμερό τους όλο και αυξάνεται. Πώς θα προστατευτούν αποτελεσματικά οι ανήλικοι αυτοί. Ευχαριστώ, Κατρίνα. Η κυρία Λόριστον. Thank πάρα πολύ, Κλοντ, και συγχαρητήρια, κυρία Γιώργα. Ευχαριστώ και για την προτεραιότητα που δώσατε σε ζητήματα προστασίας δεδομένων και εφαρμογής. Έχουν απομείνει 15 μήνες για να οριστικοποιηθεί η διαδικασία. Και θυμάστε πως όταν προετοιμάζαμε τον ε, κανονισμό ένα από τα ζητήματα αυτά που μας απασχολούσε με τα κράτη-μέλη στο διάλογο ήταν το ζήτημα των ε, αρμοδίων για την προστασία δεδομένων. Η ε, οδηγία έλεγε πως θα έπρεπε να είναι στις διοκτικές αρχές ε, ή στις επιχειρήσεις. τι θα γίνει τελικά, γιατί απαιτείται προετοιμασία, εκπαίδευση και ζήτημα πειθαρχίας, γιατί εξ όσων γνωρίζω η εκπαίδευση δεν ε, περιλαμβάνεται στην διδακτική ύλη, στις νομικές σχολές, σε άλλες σχολές, οπότε δεν υπάρχει κάποιος ειδικό. Οπότε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορέσουμε σε 15 μήνες να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Σας ευχαριστώ, Μπόνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίαση και ευχαριστώ και συγχαρητήρια Κλοντ για την εκλογή σας. Νομίζω πως θα είναι θετική για την Επιτροπή μας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα ο κώδικας συμπεριφοράς για την καταπολέμηση του μίσου στο διαδικτύο. Στο διαδικτύο. Οριστικοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες. Έχει γίνει μια πρώτη αξιολόγηση από την Κομισιόν. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια, προβλήματα για την πλήρη εφαρμογή του κώδικα αυτού, ειδικά στο εθνικό επίπεδο οργανώνω την Παρασκευή, την σχετική διάσκεψη στην Βαρσοβία. Έχω προσκαλέσει και εκπροσώπους της Κομισιόν ε, και είναι σημαντικό να δούμε τι γίνεται στο εθνικό επίπεδο. Σκοπεύει η Κομισιόν ε, να κάνει κάποιες άλλες δραστηριότητες, να αναλάβει άλλες δραστηριότητες στον τομέα Κατόπιν, εφαρμογή της οδηγίας για τη κριτική μεταχείριση Έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές από την ομάδα του άρθρου 29 και ε, βεβαίως άλλα είναι έτοιμα για το 2017. Χρειάζεται λοιπόν να επιταχυνθεί η δουλειά μας στον τομέα αυτών. Τι ε, μπορούμε να κάνουμε. για να υπάρξει ακριβώς η εναρμόνιση στον τομέα αυτόν. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Κυρία Επίτροπε, είπατε ότι θέλετε να διατηρηθεί αυτή η φιλοδοξία για την οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος η οποία δεν αφορά μόνο το ξέπλυμα χρήματος, αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τι μπορείτε να μας πείτε λοιπόν, ποια προβλήματα αναμένατε όχι από το Κοινοβούλιο μάλλον, αλλά από τις κυβερνήσεις για τις ε, προτάσεις σας. Για ζητήματα δηλαδή διαφάνειας ως προς τον τελικό δικαιούχο και αν θα επανέλθουμε στο φυσικό πρόσωπο και να φύγουμε από το παραθυράκι που είχε η πρώτη οδηγία που επιτρέπει να σταματήσει η ταυτοποίηση στον διαχειριστή και κατόπιν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί εάν συνεχίζουμε να επιτρέπουμε σε ένα κράτος μέλος να προχωράει σε νόμιμο ξέπλυμα χρήματος που λέγονται οι χρυσές βίζες πάτε στο σχετικό site της Προεδρίας της ε, Μάλτας και υπάρχει βλέπετε εκεί πέρα no more taxes και τα λοιπά site που προσπαθούν να προσελκύσουν άτομα μεγάλου πλούτου για να ξεπλύνουν τα χρήματα στη χώρα και να αποκτήσουν υπηκότητα. Μπορούμε να συνεχίσουμε να το επιτρέπουμε αυτό. Χωρίς κάποια έρευνα. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να γίνει μια φορολογική έρευνα. Δεν διασφαλίζεται καμία δέουσα επιμέλεια από οποιονδήποτε ενδιάμεσο στην διαδικασία αυτή της χρυσή θεώρησης. Σας ευχαριστώ. Ποιος Vielen ähm, äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω αρκετέ ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα για την Συμφωνία Ομπρέλα. Χαίρομαι που έχει φτάσει ε, εκεί που έχει φτάσει στην ε, Αμερικανική νομοθετική διαδικασία. Όσον αφορά τώρα τις προϋπάρχουσες ε, αποφάσεις για την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα θα έχουμε τα ίδια προβλήματα για τα ζητήματα ασφαλείας. Για την απορρόφηση, ας πούμε, των δεδομένων. Δεύτερη ερώτηση αφορά την αντίδραση της Κομισιόν για την συμπεριφορά των βελγικών αρχών που θα βάλουν δεδομένα πιενάρια τα τρένα, δεδομένα επιβατών τρένων. τρίτη ερώτηση. Την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω υπήρξε μια ανακοίνωση ή μια δήλωση στον τύπο για το TFTP και το PNR και υπήρχαν κάποια προβλήματα που διαπιστώθηκαν. Τι κάνουμε τώρα με τα προβλήματα αυτά. γιατί φαίνος είχαν το πρόβλημα ότι υπήρχαν πολλοί εργαζόμενοι που είχαν πρόσβαση στα δεδομένα και αφετέρου ε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα ποια κράτη μέλη συμμετέχουν και ποια όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι ε, θα συμβεί όταν υπάρχουν πολλές αξιόπινες πράξεις ενός ατόμου που αφορούν και τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητας μεταξύ άλλων. Πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά εδώ τις αρμοδιότητες και πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κιέγγε, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Κλοντ. Ευχαριστώ την, σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, την καταπολέμηση του hate speech, του λόγου μίσους. Μιλήσατε για τη συμφωνία που έγινε. Με το Google, YouTube, Facebook, Twitter. Δεν νομίζετε ότι πρέπει να έχουμε και μία προσέγγιση νομοθετική για να καταπολεμήσουμε αυτές τις ομιλίες μίσους. Τι πρόθεση έχει η Κομισιόν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, πώς θα αντιμετωπίσει. Σήμερα, εκτός από αυτές τις ομιλίες, ε, στο διαδίκτυο έχουμε και ψευδείς ειδήσει. Ε, τι σκοπεύει να κάνει στο μέλλον η Κομισιόν για να αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα. Δεύτερον, για την εθνική στρατηγική καταπολέμηση της της φοβίας ε, των, ανθρω... ανθρώπων. Συνδέεται με την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Για να έχουμε μια καλή στρατηγική θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλες τις άλλες διακρίσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, επιστρέφω σε αυτού του είδους την φοβία ε, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ετοιμάζει ένα εγχειρίδιο καλών πρακτικών με βάση τα όσα κάνει ας πούμε η Ολλανδία, η οποία έχει μια τέτοια στρατηγική. Την καταπολέμηση λοιπόν ε, αυτής της φοβίας, ε, του hate speech, αυτά για να αντιμετωπίσουμε δεν θα πρέπει να προβλέψουμε μόνο τις κυρώσεις, αλλά και την εκπαίδευση ε, των ανθρώπων και την εκπαίδευση ψηφιακή. Αλλά και αντίθετα άλλου τύπου αφηγήματα, α πούμε, εναλλακτικέ λύσεις. Τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει την αφροφοβία. κυρια uh, Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τη δέσμευσή σας και για την ε, διαθεσιμότητά σας. Έχω μερικά θέματα. Καταρχήν, ε, Σύμβαση Κωνσταντινούπολη για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Το Νοέμβριο θετήσαμε σχετικό ψήφισμα και οργανώσαμε και ακρόαση. Και εκεί ρωτήσαμε σε τι φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσει με τα κράτη-μέλη προκειμένου να προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ξέρω ότι ασχολείστε με αυτά τα θέματα. Ε, το συζητήσατε με τη Μαλτέζικη Προεδρία και πού βρισκόμαστε και μάλιστα ως συνεισηγήτρια για την συνθήκη, για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ασχοληθήκαμε με, τις, με τους ενδιασμούς που έχουν κάποιες ε, χώρες ό,τι αφορά την, τον ορισμό και το καθεστώς της έννοιας του φύλου, το gender, γιατί μιλάμε για ε, βία λόγου φύλου. Και μάλιστα η σύμβαση προβλέπει ότι η βία ε, για λόγους φύλου στοχεύει εις βάρος των γυναικών μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες, λόγω του φύλου τους. Θα ήθελα πάντως να ε, επαναλάβουμε την έκκληση για επανάληψη του διαλόγου με τα κράτη-μέλη που έχουν ενδιασμού για το θέμα αυτό, σε συνδυασμό και συντονισμό με το Συμβούλιο της Ευρώπης, που φέρει και την πρωταρχική ευθύνη για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολεως. Δεύτερο ζήτημα, η στενοποίη, τα διέξοδα, ε, δύο είναι τα βασικά διέξοδα, ε, η οδηγία κατά των διακρίσεων το θέμα της ίσης μεταχείρισης και των ίσων δικαιωμάτων που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που άπτεται των οικουμενικών μας αξιών. Θα πρέπει λοιπόν να προωθηθούν οι διαπραγματεύσεις και να ξεπεράσουμε επιτέλους αυτό το, αυτό το σκόπελο του κόστους. Ένα αντίστοιχο θέμα και αδιέξοδο, το θέμα της πρόσβασης του κοινού ε, στα ε, έγγραφα. Και εκεί έχει κολλήσει το θέμα εδώ και πολύ καιρό στο Συμβούλιο. Θέλουμε να ενισχυθεί η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα έγγραφα των ε, κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Και επίση το ζήτημα των παιδιών. Ξέρω ότι σα ενδιαφέρει αυτό το θέμα, αλλά ο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων δυστυχώ δεν έλαβε υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών. Απέτυχε στο θέμα αυτό και έχει πολύ κατακαιρματισμένη προσέγγιση. Και η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι απαράδεκτη. Και τέλος, μόλις υπευλήθη η πρόταση για την αξιολόγηση της οδηγίας ό,τι αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών. Ελπίζω να είστε πιο φιλόδοξοι, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ανεπαρκής αυτή η αξιολόγηση που έγινε. Ευχαριστώ κύριο Μάρεκ Γιούρεκ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και συγχαίρω θερμά τον Κλοντ για την επανακλογή του και για το δεύτερο αυτό μισό της κοινοβουλευτικής θητείας. Θα ήθελα να αναφερθώ στα θέματα των διακρίσεων. Η Επίτροπος, στην τελευταία συζήτηση που έγινε για την Πολωνία, στο Κοινοβούλιο, εκφράσεται κάποια κατανόηση για εκείνους ε, που τάσσονται υπέρ της ε, νομιμότητας των αυλώσεων δεν θα συζητήσουμε εδώ τις διαφορετικές θέσεις, ε, ούτε την κατανόηση που δείξατε για αυτή την πλευρά. Ε, εγώ θα επικεντρωθώ στη νομική πτυχή. Πολλές ε, χώρες μέλη, η Πολωνία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Σλοβακία, έχουν επιβεώσει νομοθετικά τα ανθρώπινα δικαιώματα του παιδιού πριν τη γέννηση, πριν τον τοκετό. Και μάλιστα έχουμε και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην περίπτωση της υπόθεσης Μπρίσλε κατά της Greenpeace. Εκεί η απόφαση του δικαστηρίου μιλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όχι αμέσως πριν την, το τοκετό, αλλά και σε φάση, στη φάση την εμβρυϊκή, στην εμβρυϊκή φάση της ζωής. Αυτό το αναγνώρισε και η νομολογία του ΔΕΚ, λοιπόν. Θεωρώ, λοιπόν, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι κοινοτικό θεσμικό όργανο και μάλιστα που οφείλει να εξυπηρετεί και να εργάζεται υπέρ τη συνεργασία, θα πρέπει να λάβει υπόψη και αυτά τα νομικά επιχειρήματα και αυτή την νομοθετική κατάσταση. Γιατί εκτός της νομολογίας έχουμε και το κράτος δικαίου και τη νομοθετική κατάσταση των κρατών μελών. Γιατί πολλές φορές κάνετε επίκληση του κράτους δικαίου και παρόλα αυτά δεν τα τηρείτε. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που ε, επικαλείται τα, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να ξεχνάω ότι η ζωή είναι θεμελιώδης δικαίωμα, άσχετα με το αν θα δεχτούν διακρίσεις ε, εις βάρος των μη γεννηθέντων παιδιών, εις βάρος των ευρείων. Θα πρέπει λοιπόν ε, να δούμε πώς αντιμετωπίζονται οι παράνομες ενέργειες, γιατί μερικές φορές παράνομα εφαρμόζονται τέτοια δικαιώματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά την θέση της Πολωνίας ε, για το θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής. Αναφέρθηκε η δημοσιονομική πίστη που θα σκεφτεί στην Πολωνία προκειμένου να απάδει από τις συνταγματικές της αρχές. Και μάλιστα ε, ζητά ε, πολλέ φορέ επικριτέ τη Πολωνία μα ζητούν να εμείνουμε σταθερά στις συνταγματικέ αρχές. Τώρα, πώ ξαφνικά θέλετε να αποκλίνουμε από τις συνταγματικέ αρχές μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της συμμετοχή στην εισαγγελική αρχή. Ευχαριστώ οι δύο τελευταίοι ομιλητές μας και σας θέρμο παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το ένα-δύο λεπτά για να έχουμε χρόνο και για τις απαντήσεις από την Επίτροπο. Ο κύριος Τσάκη. Σας ευχαριστώ. Θα μιλήσω στην δική σας μητρική γλώσσα που τη χάνει να την ομιλώ και εγώ για να συνεννοηθούμε καλύτερα. το Συμβούλιο ασχολήθηκε με διάφορα θέματα που βρίσκονται σε διέξοδο, αλλά πότε θα έχουμε επιτέλους κάποια έγγραφα. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, σύντομα. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας Κάθε επιτυχία εύχομαι. Στην κυρία Γιώργα. Δύο ανησυχίες έχω. Που βασίζονται σε πράγματα τα οποία ήδη έχουν συζητηθεί από τους συνοδελφούς. Πρώτα απ' όλα το μέλλον του ποινικού δικαίου για τις ε, δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ε, η διαδικασία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Για να συμβεί επιτέλους κάτι τέτοιο, θα ήθελα να κάνετε μία δήλωση για την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί επιτέλους. Δεδομένου του ότι έχουμε αρκετό περιθώριο για συμβιβασμούς μέσω της ε, οδηγίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσει επιτέλους αρμοδιότητες ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά την προστασία δεδομένων ε, και την συμφωνία Ομπρέλα. Περιέχει την ε, σχετική νομοθεσία των ΙΠΑ ε, για την δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και για Ευρωπαίους πολίτες επιτέλους για να μπορούν να προσφύγουν με βάση τις Αμερικανικές προδιαγραφές προστασίας δεδομένων. Θα ήθελα λοιπόν να αξιολογήσετε τις δυσκολίες ε, που μπορεί να προκύψουν δεδομένης της αλλαγής Αμερικανικής κυβέρνησης. για την ισοτιμία της σχέσης ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ευχαριστώ συνάδελφοι, καλύψατε νομίζω τα σημαντικότερα ζητήματα και εντός του χρόνου. Και τώρα τουλάχιστον έχει λίγο χρόνο να απαντήσει η Επίτροπος για ε, τις πάρα πολλές ερωτήσεις με ευρύτατη θεματολογία. Έτσι είναι τα πράγματα πάντα Οπότε έχετε τον λόγο. Και σας παρακαλώ αναφερθείτε και στην ερώτηση της κυρίας Σίνετφελτ. Ναι, ναι. Νομίζω έχουμε μέχρι τις 6.30 ο πρόεδρος. Ναι, κοιτάξτε. Αν επιλέξουμε ένα-δύο μεγάλα θέματα για τον επόμενο γύρο, ευχαρίστως να έρθω και να τα συζητήσουμε για το θέμα του PNR και την εξαίρεση. Θα αναφερθώ στο ότι μου έχουν ετοιμάσει εδώ πέρα. Άρθρο 19.1 της Συμφωνίας Ομπρέλας επιβάλλει υποχρέωση της ΗΠΑ να δώσουν στους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήρια ε, και όταν μιλάμε για δεδομένα επιβατών. Για ε, τις 17 Ιανουαρίου μας κοινοποίησαν οι ΙΠΑ ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της εσωτερικής ασφαλείας, δηλαδή τελωνία και προστασία συνόρων, θα πρέπει να συμμορφωθούν. Εάν δεν συμμορφωθούν οι ΙΠΑ, στην πράξη θα παραβιάζουν την συμφωνία ομπρέλα, κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει λόγο διακοπής τη ισχύω τη σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1. Αυτό, καθαρά νομική απάντηση. Νομικιστική, να μην πω. Δεν ξέρω, θεωρούσατε ότι τα PNR θα είχαν εξαρθεί. Μα όχι από την νομοθεσία, το νόμο περί δικαστικής προσφυγής. Για τα ένδικα μέσα μας είχατε πει πως για να, ισχύουν, να ισχύσουν αυτά οι εξαιρέσεις από το PNR και το TFTP ε, από την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων που αυτή τη στιγμή δεν τα καλύπτει θα πρέπει οι εξαιρέσεις να καταργηθούν. Δηλαδή, εκτός εάν η ε, νομοθεσία καλύπτει και το PNR και το TFTP, δεν ισχύει η συμφωνία και το έχετε επιβεβαιώσει εσείς και η υπηρεσία σας. Δεν έχουν ανακληθεί λοιπόν οι εξαιρεσει ε, και ούτε επί Προέδρου Ομπάμα δεν είχαμε καμία ένδειξη ότι θα ανακληθούν. Οπότε, εάν η συμφωνία είναι να τεθεί ενισχύ την 1η Ιανουαρίου και δεν έχουν ανακληθεί εξαιρέσει, δεν μπορεί να ισχύει. Δεν θέλω να μπω σε ε, στις νομικές πτυχές. Έχω το κείμενο εδώ πέρα και τα επιχειρήματα μπροστά μου. να σας τα στείλω γραπτός, να σας στείλω μία απάντηση για να καλύψω όλο το πλαίσιο. Για να επανέλθω στο θέμα της μετανάστευσης αύριο, ε, θα έχετε εδώ τον κύριο Βραμόπουλο και θα καλύψετε το θέμα. Ξέρω πως ρωτήσατε συγκεκριμένα για τα γυναικόπαιδα. Ε, η κυρία Κορατσαμπίλτ έφυγε. Ναι. Είπατε ότι δεν θέλετε μία γενική απάντηση. Αλλά αυτή είναι η απάντηση. Εστιάζουμε στην δημιουργία ουσιαστικών δίκλειδων ασφαλείας ε, στη διαδικασία σύλλου στα γυναικόπαιδα, γιατί είναι ευπαθείς ομάδες. Οπότε όταν μιλάμε για γυναικόπαιδα, ε, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να δημιουργηθούν ασφαλείς ζώνες όπου δεν θα κινδυνεύουν από εγκληματικότητα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα όπου συγκεντρώνονται άνθρωποι δυστυχώς. Και αν θυμάμαι καλά, οι διαδικασίες ε, ασύλου απαιτούν και ειδικέ συνθήκες για τις ε, συνεντεύξεις με γυναικόπαιδα που έρχονται στις ζώνες υποδοχής και ειδική μεταχείριση για να είναι ασφαλής ε, και να μην υποφέρουν και τους δημιουργηθεί περαιτέρω ψυχολογικό τραύμα γιατί προέρχονται ήδη από δύσκολες καταστάσεις. Επίσης, προσπαθούμε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να βοηθήσουμε την ένταξη των γυναικών στην κοινωνία. Είμαστε λοιπόν σε επαφή με τα κράτη-μέλη που ξεκίνησαν τη διαδικασία ένταξης, ε, όχι μόνο των γυναικών, αλλά και των ασυνόδευτων ανηλίκων γιατί ε, τα παιδιά που έρχονται χωρίς γονείς στην Ευρώπη θα σας δώσω ένα νούμερο από την Ελλάδα 80% των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι μεταξύ 15 και 18 που απαιτούν ειδική μεταχείριση αλλιώς ε, ε, όχι μόνο δηλαδή τροφή και στέγη πρέπει να έχουν και μία προοπτική και πρέπει οι υπηρεσίες ε, να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν προσόντα ε, και μια φυσιολογική ζωή σε κάποιο κράτος μέλος. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Αυστρία σε ένα κέντρο υποδοχής. Πραγματικά ε, χάρηκα ιδιαίτερα από τα όσα γίνονται εκεί πέρα για τα παιδιά. Όχι μόνο οι άνθρωποι στις υπηρεσίες, οι άνθρωποι της πόλης κάνουν πολλά πράγματα, οι ηλικιωμένοι βοηθάνε τα παιδιά να ενσωματωθούν. Ε, ξέρω ότι έχετε και άλλα πράγματα. Επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα έχουμε μια αποκεντρωμένη δομή. Το κείμενο έχει οριστικοποιηθεί. Θα πρέπει να απορρίψω αυτή την απεσιοδοξία. Είναι λάθος. Έχουμε οριστικοποιήσει το κείμενο. υπάρχουν σοβαρές ε, ε, και ισορροπημένες αρμοδιότητες ανάμεσα στο κεντρικό γραφείο και στο κράτος μέλος. Βασιζόμαστε ε, στους Ευρωπαίους βοηθούς εισαγγελέων και επιπλέον έχουμε καλά δεδομένα σε σχέση ωφελίας, ας πούμε, σε σχέση με το κόστος. Και όταν το ΦΠΑ ενταχθεί στις αρμοδιότητες του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία θα επιστρέψουν ε, και στον Ευρωπαϊκό Κορβανά και στους Εθνικούς Κορβανάδες. Ε, τι σχέση έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Προβλέπουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ε, προβλεπόταν ήδη στη συνθήκη της Λισαβόνας ως το γραφείο του Εισαγγελέα που θα έχει απο, αρμοδιότητες να παίρνει αποφάσεις για να διώξει και να οριστικοποιήσει ε, υποθέσεις σε προδικαστικό επίπεδο και να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, να προστατεύσει το ενωσιακό προϋπολογισμό. Αυτό το οφείλουμε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους, ειδικά στα κράτη-μέλη που είναι καθαροί εισφορείς, ναι, καθαροί συνδρομητές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτή είναι η έντονη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον ενωσιακό προϋπολογισμό. Θα υποβάλουμε μία πρόταση επίσης κανονισμού στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης τον Ιούνιο για το, για το σύστημα που θα καλύψει και ε, υπηκόους ε, τρίτων χωρών, το ΑΚΡΙΣ, και το ΑΚΡΙΣ θα πρέπει να έχει και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι, πρόκειται για μια μαζική συλλογή δεδομένων προσώπων και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για να διευθετηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. αυτό, για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε τον κανονισμό και πρέπει να γίνει αυτό σύντομα και σωστά. Τον Ιούνιο λοιπόν το Σώμα των Επιτρόπων θα υιοθετήσει το κείμενο αυτό. Υπάρχει συμφωνία με την Εστονική Προεδρία ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία της υιοθέτησης στο Συμβούλιο του κειμένου αυτού. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τη θέση όλων των κρατών μελών. Μάλιστα. Για το κώδικα ε, διοντολογίας. Άκουσα διάφορες ερωτήσεις που είναι τα εμπόδια, που είναι τα προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα ποιο είναι. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Να ξεκαθαρίσουμε στο κοινό, στους Ευρωπαίους, ότι αυτό που κάνουμε με τον κώδικα διοντολογίας είναι να αποσύρουμε τα... να σταματήσουν πια αυτές οι ρητορικέ μίσους. Οτιδήποτε λέγεται και είναι παράνομο, πρέπει να σταματήσει. Να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του φράχτη, ας πούμε. Ας πούμε, αν γραφτεί κάτι παράνομο, ας σε ένα τείχο θα πρέπει να έρθει η αστυνομία και να σβήσει αυτά, αυτά τα συνθήματα μίσους, ας πούμε. Φυσικά, αν κάτι ανάλογο γραφτεί στο ίντερνετ, φυσικά ε, εντυπώνεται πολύ περισσότερο στα μυαλά των ανθρώπων. Αμέσω, ας πούμε, υπάρχει απάντηση κτλ. Η κινητοποίηση. Εάν θέλουμε, λοιπόν, να επανέλθουμε σε αυτή τη συμφωνία των τον κώδικα διοντολογίας με τους παρόχους της προφορικής, πρέπει να καταλάβουμε ποιο δίκαιο εφαρμόζεται τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για παράνομες ρητορικέ μίσους. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να περιστήλουμε την ελευθερία λόγου. Μετά την πρώτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας, πού είναι τα εμπόδια τώρα, αυτό ήταν μια από τις ερωτήσεις. Υπάρχει έλλειψη δυναμικού. Δεν, ξέρουμε, δεν υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που γνωρίζουν, γνωρίζουν τις γλώσσες. Σε ορισμένε περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι νομικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα ορίσουν το τι είναι παράνομη ρητορία μίσους. Τι πρέπει να διαγραφεί, τι πρέπει να εξαφανιστεί και τι μπορεί να παραμείνει. Και αυτό συνδέεται πάρα πολύ καλά ε, με την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη και την ομολογία τους, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, τα ευρωπαϊκά συνταγματικά δικαστήρια καθορίζουν τι είναι παράνομη και τι νόμιμη ρητορία και τι είναι παράνομη ρητορία μίσους. Επίσης, τις κινητοποίησεις από επίσημους φορείς φυσικά τις παίρνουμε πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο σοβαρά από τις ε, γνωστοποίησεις από απλούς πολίτες η ΜΚΟ. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό την άνοιξη φέτος, να αξιολογήσουμε αν τελικά έχει σημειωθεί πρόοδος με το θέμα του κώδικα διοντολογίας. Φυσικά, Οτιδήποτε γράφεται δεν είναι ρητορία λόγου, έτσι. Εγώ πιέζω και τους παρόχους ε, πληροφορικής να είναι διαφανείς, να ενημερώνουν το κοινό για αυτό που κάνουν σε αυτόν τον τομέα, τι κατεβάζουν ας πούμε, γιατί υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα σε ρητορίε μίσους και σε απόψεις που πρέπει να προστατευθούν ε, και να εκφράζονται λόγω της ελευθερίας λόγου που έχουμε εδώ. εφαρμογή του GDPR. Πρέπει να διευκολύνουμε την εφαρμογή του κανονισμού GDPR σε όλα τα κράτη-μέλη, Το κανονισμό την, για την προστασία των δεδομένων. ο κανονισμό φυσικά είναι άμεσα εφαρμοστέως. Είναι κανονισμός σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, είναι γενικός κανονισμός και όχι οδηγία. Θα απαιτηθούν πολλές αλλαγές τη εθνική νομοθεσία, στα κράτη-μέλη, ειδικά στα κράτη-μέλη που δεν συνδέονται και δεν προστατεύουν άμεσα την, τα δεδομένα. Παραδείγματο χάρη στην εργατική νομοθεσία κτλ. Λοιπόν, τι κάνουμε για την εφαρμογή. Εστιάζουμε σε τέσσερα πράγματα. Είμαστε σε έντονες επαφές με, το, με την ομάδα εργασίας 29 που ετοιμάζει τη δράση. Αυτοί θα εφαρμόσουν αυτό το κανονισμό. Θέλουμε οι κανόνες να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κρατη Και ξέρετε ότι στο Γενικό Κανονισμό υπάρχει μια διακριτική ελευθερία, ας πούμε, ένα περιθώριο στα κράτη-μέλη. Ας πούμε, οι κυρώσεις Θέλουμε όμως να εφαρμοστούμε τον ίδιο τρόπο. Δεν θα πρέπει στη Γερμανία, ας πούμε, να έχουμε υψηλότερε ή χαμηλότερε κυρώσει από ό,τι στη χώρα μου ή στην Πολωνία, Φερρυπίν. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό επηρεάζεται και από το επίπεδο πολιτισμού, από την νοοτροπία της κάθε χώρας από τη σημασία που δίνεται στην προστασία ιδιωτικών και προσωπικών δεδομένων. Και φυσικά υπάρχουν διαφορές από κράτο σε κράτος. Αυτό είναι λοιπόν το ένα στοιχείο. Και θα σεβαστούμε απόλυτα την εξαρτησία των ε, ε, εθνικών εποπτών προστασίας δεδομένων. Τώρα, για την τροποποίηση της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, την, πάνω, την αλλαγή. Παρακολουθούμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που είναι ας πούμε, μπροστά σε αυτόν τον τομέα, π.χ. Γερμανία. Και θέλουμε να δούμε ποιε είναι οι ανάγκες στα κράτη-μέλη, τα οποία πρέπει να προβούν σε αλλαγή τη νομοθεσία και έχουμε υποσχεθεί σε αυτά να οργανώσουμε κανάλια ανταλλαγής πληροφοριών και να εξασφαλίσουμε συντονισμό εμεί από πλευρά Κομισιόν. Τρίτο πράγμα που κάνουμε για τον κανονισμό αυτό, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ε, σαφέστατοι κανόνες, ε, μονοσήμαντα ερμηνεύσιμοι για τις ε, εταιρείε και κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείε. καθαροί κανόνες για τους υπευθύνους προστασίας δεδομένων. Το ζητήσατε πολύ από εσά. Το επιβεβαιώνω. Ναι, αυτό θα είναι βασικό θέμα. Ε, επίσης, τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι αρχές προστασίας δεδομένων. Μας στέλνουν ήδη μηνύματα σως, γιατί όσους καλούς υπαλλήλου έχουν, ας πούμε, τους παίρνουν οι ιδιωτικές εταιρείες. Και υπάρχει πρόβλημα εδώ. Με δημοσίους λειτουργούς που είναι καλοί, που να είναι καλοί. Υπάρχουν κάποια ανησυχητικά νέα ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσλάβουν στην Τσεχία, α πούμε, 35.000 νέους δημοσιου υπαλλήλου για τους δημόσιου φορείς προστασίας δεδομένων. Έτσι λέει η κυκλοφορία, α πούμε. Εγώ εξήγησα στον κόσμο. Μην, μην λέτε σαχλαμάρες. Θα προετοιμάσουμε τους σημερινού σημερινούς υπαλλήλου που δουλεύουν σε, στους τομείς α, ανθρωπίνων πόρων ή σε συναφείς, ας πούμε, ε, συναφή τμήματα, δεν χρειάζεται να προσλάβετε 35.000 νέου δημοσίου υπαλλήλου, δεν αναγκάζει η Κομισιόν κανένα κρατό μέλο να προσλάβει ένα στρατό, μια τέτοια στρατιά υπαλλήλων μόνο και μόνο για να κάνουν αυτή τη δουλειά προστασία δεδομένων. Επομένω. πολλές παρεξηγήσεις θα κυκλοφορήσουν και εμείς πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά του ε, επόπτε προστασία δεδομένων και τους ε, υπαλλήλους, ε, του υπεύθυνου, Ήδη οι επόπτε έχουν εκδώσει κάποιε κατευθυντήριε γραμμές για το ποια θα πρέπει να είναι τα καθήκοντα αυτών των ειδικών υπαλλήλων για την προστασία των δεδομένων και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εξηγούμε τα πράγματα στι εταιρείε για να μην πανικοβληθούν και να μην παρασυρθούν από ιστερική κινδυνολογία, κάτι που συνέβη σε κάποια κρατημέρια. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, θέλουμε να δημιουργήσει συνθήκε ισότιμου ανταγωνισμού και καλέ προποθέσει για τι εταιρείε, ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσει να ε, τηρήσουν τι υποχρεώσει του και να μην ε, υπερφορτωθούν από νέε γραφειοκρατικέ διοικητικέ διατυπώσει. Και αυτό είναι το, το τρίτο στόχος και ο τέταρτος είναι η εκστρατεία για να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, ε, για να κατανοήσουν ε, τα νέα δικαιώματα που τους ε, κατοχυρώνει ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και να ετοιμαστούν για αυτά. Αυτή η εκστρατεία λοιπόν θα πάρει αρκετούς μήνες και θα ξεκινήσει μάλλον στις αρχές του 2018. Και φυσικά αυτό είναι και έργο των κρατών μελών, των επιχειρήσεων, των εποπτών προστασίας δεδομένων και συνεργασία όλων αυτών των φορέων. Πάντως πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αν είμαστε συστηματικοί στην προσέγγιση μας και δεν υποτιμήσουμε τα επιμέρους στοιχεία που προβλέπει ο κανονισμός, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σε ό,τι αφορά τις δικονομικές εγγύησεις ε, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, εμείς βάλαμε τα δυνατά μας και προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλες τις οικονομικές ασφαλιστικές δεκλίδες που ήδη έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβλέπεται και η νομική συνδρομή που πρόσφατα υιοθετήθηκε και είναι το τελευταίο στοιχείο, το πιο πρόσφατο. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δράσεις των δικηγόρων που προετοιμάζονται, γιατί και αυτή τη δουλειά τους κάνουν, οι συνηγοροί περάσπισης, Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε παραθυράκια στις προτάσεις και αβεβαιότητες ή, ανα... ή ασάφειες ως προς, την... Ε, ως προς τον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, γιατί θα είναι πολύ εύκολο στόχος αυτή η νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή, δεν θα πρέπει να υπάρχουν κενά λοιπόν. Και Επίσης και για τους υπόπτους θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις ε, ύψιστες ε, ε, δικονομικές εγγύσεις. Γιατί για φανταστείτε να σας κατηγορεί κάποιος για διαφθορά ή για απάτη ενώ είστε αθώος. Δεν θα πρέπει να μπορεί κανείς να σας εγκλωβίζει σε αυτό το σημαντικό ε, διεθνές όργανο σε μία χρονοβόρα ε, έρευνα που μπορεί να κρατήσει και 5 και 10 χρόνια. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να αποτραπεί οπωσδήποτε να προστατευτούν και τα δικαιώματα των υπόπτων. Αυτά. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα κέριο. Α, ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι έτοιμη για την επιστολή που ανακοινώσατε και θα κάνω ό,τι μπορώ. Ε, θα χρησιμοποιήσω όλες τις αρμοδιότητες που έχω για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση του αριθμού κλίση 116 γιατί είναι σημαντικό στοιχείο του συστήματος η διασφάλιση αυτής της γραμμής. Το σημαντικό είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό υποστηρίζουμε. Σύσσωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως στην Επιτροπή μας είμαστε υπέρ της συνεργασίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Όποιο σύστημα και αν έχουμε, να εξασφαλιστεί συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, και η δική μου μία μικρή συμπληρωματική ερώτηση, συγγνώμη. Ναι, ξέπλυμα χρήματο, νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Κύριε Αγκόμε, ποιο είναι το μείζον πρόβλημα, τα δημόσια μητρώα. Και με ενοχλεί η θέση των κρατών μελών Καταλαβαίνω βέβαια τα επιχειρήματά τους ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα και του δικαιώματος ε, του κοινού να γνωρίζει τα πράγματα. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να δούμε τι είδους δεδομένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά τα δημόσια μητρώα. Και τότε όταν έχουμε όνομα, εθνικότητα, κατάσταση επιχειρήσεων, κάτι που να μην θέτει σε κίνδυνο κανέναν. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει που δεν είναι να θέτουν σε κίνδυνο οποιονδήποτε. Και τώρα υπάρχουν πιέσεις για να μην είναι πλήρως προσιτό στο δημόσιο αυτό το μητρό, τα δημόσια αυτά, να μην είναι δημόσια τελείως αυτά τα μητρώα και νομίζω ότι οι εξελίξεις έχουν γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά είμαι συνέχεια σε εκνευρισμό και γιατί αυτά τα μέτρα που στόχο έχουν την αποτροπή τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία έχουν και αυτά κολλήσει, έχουν μπλοκαριστεί γιατί ε, εμπεριέχονται στην ε, γενικότερη αυτή νομοθεσία και έχει αποτελματωθεί κατάσταση και ω προ αυτά και αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερω. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη να δεχτούν τα δημόσια μητρώα. Και δεν ξέρω προς τι όλη αυτή η αντίσταση και η διαμαρτυρία, γιατί στην τέταρτη εκδοχή τι οδηγίε για την καταπολέμηση τη νομοποίηση χρημάτων από παράνομε δραστηριότητε, υπήρχε επιλογή είτε πλήρω δημόσια, μητρό, είτε για ορισμένου φορεί μόνο. Και κάποιε χώρε ήδη προτίμησαν τα πλήρω δημόσια μητρό και τελικά τίποτα κακό δεν έγινε. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω την αντίσταση των, υπόλοιπων κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγής και του φορολογικού παραδείσου, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία θα πρέπει απλώς να εφαρμόσουμε σωστά την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτό είναι που ε, μας λείπει. Ευχαριστώ τους Δερμηνείς για την υπέρβαση. Ζητώ συγγνώμη και εγώ το ίδιο. Ζητώ συγγνώμη, λέει η Επίτροπος. Σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές για την καταπολέμηση της ρητορική του μίσους, έχουμε την απόφαση πλαίσιο κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. που κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγες την κατάσταση στα κράτη-μέλη και να τα πιέζουμε να εφαρμόσουν σωστά αυτή την απόφαση πλαίσιο. Μέχρι στιγμής μόνο τα μισά κράτη έχουν εφαρμόσει την ε, οδηγία πλαίσιο πλήρως, ενώ τα υπόλοιπα δεν το έχουν κάνει. Γι' αυτό και θα το ξαναεπισημάνω αυτή την εβδομάδα, ίσως την Παρασκευή, στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, αλλά και στο μέλλον και σε μεμονωμένα κράτη-μέλη, πιέζουμε για να εφαρμοστεί σωστά αυτή η οδηγία, η απόφαση πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τι ανακριβεί ψευδεί ειδήσει ή τον αντίλογο στη ρητορική του μίσου. Δεν έχουμε προγραμματίσει συγκεκριμένε δράσει. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε το δεδολογικό κώδικα για την ρητορική του μίσου. Αυτό ισχύει και για την ε, ομοφιλοφοβία ή τις επιθέσεις ε, της κατά των γυναικών, γιατί δεν είναι θέμα μόνο ρατσισμού και ξενοφοβίας, είναι ευρύτερο το φαινόμενο. Επίσης έχουμε και την πρωτοβουλία της ε, κυρίας Μογκερίνη και έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται κατά της ε, με το θέμα της φιλετικής προπαγάνδας. Και συγγνώμη, κατά της ρωσικής προπαγάνδας και προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και, το, και τις ψευδείς ειδήσει και στηρίζονται, προσπαθούν να στηριχθούν σε πραγματικά δεδομένα, σε, πραγματικά περιστατικά και στοιχεία. Δεν έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν, να κατεβάσουν οποιαδήποτε είδηση, αλλά έχουν το δικαίωμα να διερευνήσουν αυτές τις ψευδείς ειδήσει και να καταλήξουν στο συμπέρασμα και το κατά πόσο τα νέα αυτά είναι όντως ακριβή ή ανακριβή, ώστε τα διάφορα το δικό του site να φαίνει και τον αντίλογο, να δείχνει την πραγματική κατάσταση και όχι αυτοί που παρουσιάζουν αυτά τα ψευδή και ανακριβή στοιχεία. Τώρα, παρακολουθούν, δεν, δεν ασχολούνται καθόλου με άρθρα που απλώς εκφράζουν ιδέες, ε, εμένουν σε πραγματικά περιστατικά, σε πραγματικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ, ήταν πολύ λεπτομεριακές οι απαντήσεις, αλλά θέλω... Ναι, σας ευχαριστώ. Πρέπει να προγραμματίσουμε καλύτερα τις συνεδριάσεις για αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν είναι για να τα παίρνουμε έτσι ελαφρά. Αλλά χαίρομαι που αφιερώσαμε τόσο χρόνο, ειδικά για αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ κύριε Πίτροπε. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο και θα ήθελα κάποια στιγμή να πάνε και στα σπίτια του οι διερμηνείς. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ και τους βουλευτές. Ευχαριστώ που μείνατε για να απαντήσετε. Την Παρασκευή θα είστε στο Συμβούλιο, έτσι θα μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια αντίδραση ως Κοινοβούλιο, ως Επιτροπή Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε προσεχώς και σας ευχαριστώ. Συνάδελφοι, 9.45 αύριο το πρωί. Ε, τρεις ώρα χαρτί ο κύριος Αβραμόπουλος. Σας ευχαριστώ όλοι για τη συνεδρίαση.